Right, good morning everybody. Uh, Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που ήρθε και κάποιος ε, νωρίς εδώ πέρα. Συζήτησα ερχόμενη εδώ με τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και του λέω ποιος κουβαλιέται εδώ πέρα ε, στις 9 η ώρα. Και μου λέει, μα εγώ τους φέρνω όλους γιατί κάνω τις εφοριε πρωι πρωί-πρωί και μια φορά την πατήσανε και έκτοτε έρχονται. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή για τον προϋπολογισμό. Ο Άσλι Φόξ είναι ο αρμόδιος στην Επιτροπή μας. Τι προτείνω λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δώσουμε το λόγο στον Άσλι. για να μιλήσει και μετά στον κύριο Λαβίερ και μετά σε οποιονδήποτε άλλον ε, θέλει να παρέμβει. Α, κάποιοι έχουν έρθει που ξέρουν το θέμα. Οπότε ελπίζω να γίνει κάποια συζήτηση. Έχετε λοιπόν το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που είναι κατάμεστη η αίθουσα. Καλωσορίζω τον κύριο Λαβίρ. Δεν σας ζηλεύει κανείς βεβαίως, γιατί έχετε να ισορροπήσετε τα αιτήματα της Κομισιόν των Κρατών Μελών και ημών των Ευρωβουλευτών. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στις γενικές αρχές ε, του προπολογισμού, δηλαδή να πω πως θεωρώ πως ο υπερπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Νομίζω πως θα ήταν τελείως παράλογο η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει οποιαδήποτε αύξηση στις δαπάνες σε καιρό που οι φορολογούμενοι στις χώρες βλέπουν να αυξάνονται οι φόροι και να μειώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες. Όταν η Κομισιόν κάνει μάθημα σε κάποιες χώρες της Ευρωζώνης και τους λέει να κόψουν πολλές δαπάνες είναι λάθος μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Ιδεοδός θεωρώ πως πρέπει να περικοπεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι πως ε, δεν θα το στηρίξει η πλειοψηφία στην Επιτροπή ή στην Ολομέλεια. Οπότε, κύριε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε θεωρώ, είναι να παγώσετε σε πραγματικούς όρους τον προπολογισμό, δηλαδή να μην ξεπεράσετε τον πληθωρισμό. Αν και ξαναλέω πως η προτίμησή μου είναι κάπως πιο φιλόδοξη. Τώρα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής μας πολλοί βουλευτέ ε, μπορούν να λένε πως ε, χύψη ο οργανισμός πρέπει να έχει περισσότερα λεφτά για να εκπληρώσει τις απαιτήσει του ή για να ρυθμίσει καλύτερα τις τράπεζες ή τις ασφαλιστικές εταιρείε ή ό,τι κάνει. Πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος για να εξοδέψουμε ε, περισσότερα λεφτά στα διάφορα πράγματα που μα αρέσουν. Και ίσω σε κάποιε γραμμέ αρμοδιότητας της επιτροπή μας να υπάρχουν κάποια θεσμικά όργανα που αξίζουν περισσότερα λεφτά και θεωρώ πως όταν οι βουλευτές ε, κάνουν κάτι τέτοιο πρέπει αυτό να το αντισταθμίζουν με περικοπή αλλού. Δηλαδή η Επιτροπή μας δεν πρέπει να επιβαρύνει τον προπολογισμό. Αν ένα μέλος θεωρεί πως η ΕΣΜΑ χρειάζεται περισσότερα λεφτά, κάποιο άλλο πρέπει να πάρει λιγότερα. Και να έχουμε την ειλικρίνεια να εξορροπήσουμε τις αυξήσεις κάπου με περικοπές κάπου αλλού που είναι ευθύνη μας. Οπότε κύριε Λαβίρ, αυτά θα πω μόνο και... Και δεν θα επεκταθώ τώρα γιατί τους ή άλλως δεν θα έχουν και αποτέλεσμα αυτά τα οποία θα έλεγα. Σας ευχαριστώ κύριε Λαβία. Ευχαριστώ κύριε Φόξ για τα σχόλιά σας και τις συνδέξεις. Όπως ε, Γνωρίζετε, η μακρά διαδικασία του προπολογισμού ξεκίνησε με την έγκριση από την Ολομελία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των κατευθυντηριών γραμμών για τον προπολογισμό το 2013. Αυτή είναι μια μακρά διαδικασία η οποία θα μας κρατήσει απασχολημένου όλο το έτος. Εγώ ζήτησα να μπορώ να συμμετάσχω στις συνεδριάσεις όλων των επιτροπών για να έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσει όχι μόνο τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προπολογισμό, αλλά και ορισμένα στοιχεία που ίσως να είναι πιο γνωστά στα άτομα που ε, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ε, Προπολογισμού ε, και είναι και μέλη άλλων επιτροπών, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούν να γίνουν και οι σωστές αξιολογήσεις ως προς τον προπολογισμό. Βρισκόμαστε στο τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών. Ο προπολογισμό για το 2013 είναι ε, το τελευταίο έτος της περίοδου προγραμματισμού, της ε, περίοδου 2007-2013 και όπως ε, πάντοτε συμβαίνει, καθώς το ακολουθήσει το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, Περνάμε, από, περνάμε προς όλα και περισσότερες απαιτήσει πληρωμών, γιατί τα κοινοτικά προγράμματα, κυρίως αυτά που είδαμε στο πρώτο τμήμα. Είχαμε αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά κατόπιν ε, απαιτούνται πληρωμές, όπως τα προγράμματα τα περιφερειακά, τα προγράμματα έρευνας. Δηλαδή έχουμε ε, καταρχήν διαγωνισμούς, ε, στη συνέχεια ανάληψη υποχρεώσεων και στη συνέχεια πληρωμές. Και φτάσαμε στη στιγμή όπου υπάρχει ισχυρή ανάγκη, μια μεγάλη ανάγκη για πληρωμές και για όσα είπε ο κύριος Φόξ σε σχέση με τον ε, προπολογισμό της λιτότητας είναι αυτά όλα πραγματικά είναι αληθή. Πρέπει να κάνουμε ε, έναν ε, προϋπολογισμό λιτό, δηλαδή δεν πρέπει να προσθέσουμε περαιτέρω δαπάνες που να μην συνάδουν με τις προτεραιότητες, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Ευρώπη η Κομισιόν ε, ανέλαβε υποχρεώσεις ε, τα περασμένα έτη που σήμερα μεταφράζονται σε πληρωμές. Έχουμε κάποιους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσουμε και ξέρουμε πολύ καλά πως ε, οι λεγόμενες υποχρεώσεις αυτές σήμερα φτάνουν στα 200 δισεκατομμύρια. Έτσι λοιπόν, κατόπιν ε, των αναλήψεων υποχρεώσεων, ε, έχουμε τις υποχρεώσεις πληρωμών. Δεν μπορούμε να μην ε, πληρώσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε πριν κάποια χρόνια. Μπορώ λοιπόν, και να σας δώσω μία ιδέα. Θα δείξω στον συνάδελφο, αλλά μπορούν να το δουν και άλλοι, το γραφικό σχήμα όπου αναφέρονται τα αιτήματα πληρωμών από τα κράτη-μέλη το τελευταίο έτος. Στα τέλη του 2011, τον τελευταίο μήνα του 2011, το Δεκέμβριο δηλαδή, παρουσιάστηκαν από τα κράτη-μέλη νόμιμες απαιτήσει ε, πληρωμών για 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως ε, η Κομισιόν είχε στα ταμεία της μόνο 5 ε, δισεκατομμύρια για να πληρώσει. Έτσι λοιπόν ε, περίπου 10 δισεκατομμύρια πέρασαν από τον προπολογισμό του 2011 στον προπολογισμό του 2012 για πληρωμή. Και αυτό ε, μπορεί να μας οδηγήσει στο εξή να έχουμε ένα προοδευτικό κύμα ε, για απαιτήσει πληρωμών ε, που θα μετακινείται και γνωρίζουμε ότι για πολλά προγράμματα έρευνας και για ορισμένες γραμμές προπολογισμού για την περιφερειακή πολιτική οι δεσμεύσει, δηλαδή τα κονδύλια που έχουν εκταμιευτεί ε, δεν θα είναι αρκετά. Έτσι λοιπόν ζητάμε από την Επιτροπή να είναι ρεαλιστική στο προσχέδιο προπολογισμού που θα δημοσιεύσει στις 25 Απριλίου και γι' αυτό ζητήσαμε από την ε, Επιτροπή να παρουσιάσει στο δυνατόν πιο ακριβείς προβλέψεις για τις ανάγκες, την άλλη ή ανάγκη των ειδικών επιτροπών με αναφορά στις γραμμές προϋπολογισμού που αφορούν τα θέματα των διάφορων επιτροπών θα έχει ένα νόημα, θέλει να έχει ένα νόημα. Ακριβώς αυτό που είπε ο συνάδελφος Φόξ. Και το νόημα είναι το εξής. Αν έχουμε τη βούληση να ενισχύσουμε ορισμένες γραμμές προϋπολογισμού πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε και σε θέση να εντοπίσουμε και τις αρνητικές προτεραιότητες. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζητάμε περισσότερους πόρους για περισσότερες γραμμές προϋπολογισμού χωρίς να μπορούμε να ενταπίσουμε, να προσδιορίσουμε ορισμένες γραμμές που θα μπορούσαν ε, εν μέρη να περικοπούν. Έτσι λοιπόν, καλό τι επιτροπές και σήμερα την Επιτροπή ΕΚΟΝ να κάνει μια υπεύθυνη πρόβλεψη, δηλαδή μια πρόβλεψη όπου σε κάθε προτεραιότητα για την οποία θεωρούμε ότι υπάρχουν πρόσθετοι απαραίτητοι πόροι, να υπάρχει ίσως και η δυνατότητα να εντοπίσουμε και άλλες γραμμές στις οποίες μπορούν να γίνουν κάποιες περικοπές. Αυτή είναι η γενική κατεύθυνση, ακριβώς γιατί θέλουμε να έχουμε έναν υπεύθυνο και λιτό προϋπολογισμό αφενός, αλλά και αφετέρου να είναι σε θέση να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις προτεραιότητες που ψηφίσαμε. Οι προτεραιότητες που ψηφίσαμε είναι απασχόληση και ανάπτυξη και κυρίως ε, απασχόληση των νέων. Και έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τις ε, γραμμές που αφορούν τις δύο προτεραιότητες ε, γνωρίζοντας ότι ο προϋπολογισμός ε, της Ένωσης μας επιτρέπει μόνο συγκεκριμένες γραμμές κατεύθυνση σε σχέση με τις προτεραιότητες και δεν μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα με τους πόρους που μπορούμε να διαθέσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν παθιάζομαι τόσο με τα δημοσιονομικά θέματα, γιατί πολλές φορές ε, έχουμε την αίσθηση ότι ε, δεν υπάρχει συνέπεια γιατί εξηγούμε κατά θέλουμε να κάνουμε και κατόπιν βλέπουμε ότι δεν μας στάνουν τα αριθμητικά στοιχεία. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μέλο του Επιτροπή εδώ και 28 χρόνια. Ποτέ δεν ε, ε, στο Δήμο μου συμμετέχω 28 χρόνια και επανεκλέγομαι. Ποτέ δεν έχω αυξήσει του φόρου. Λοιπόν, άκουσα προτάσει ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και συνεπεί. Λοιπόν, α μην έχουμε ψευδεστήσει. Τα θέματα που συζητούμε τώρα δεν τα συζητούμε σοβαρά, γιατί ξέρουμε ότι δεν θα ληφθεί καμία απόφαση για το προπολογισμό προπολογισμού πριν να γίνουν οι γαλλικές και οι γερμανικές εκλογές. Έτσι λοιπόν, απλώς εδώ λέμε κάποια λόγια για να δικαιολογήσουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Είπατε πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ζητάτε παραπάνω. Εγώ βέβαια, πολύ ωραία, δεν θέλω να ζητήσω παραπάνω, απλώς θέλω να είμαστε συνεπείς με αυτό που ζητάμε στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε ή ε, καταυτόχρονα να βλέπουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να ζητούν να λάβει κάτι η Ευρώπη και να γράφουν επιστολές και να για να λένε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν μέχρι το 2020 ούτε επίσης ε, θα πρέπει να βασιζόμαστε σε προϋπολογισμούς που δεν είναι στη διάθεσή μας και σε σχέση με τους διερμηνείς. Ακούω παντού ότι πρέπει να μειωθούν τα έξοδα της Διερμηνείας, θα πρέπει να υπάρχει εξορθολογισμό του συστήματος και να καταργήσουμε αυτές τις δαπάνες ή να τις μειώσουμε. Και κοιτάξτε, αυτό όμω είναι κάτι αυτοκτονικό για την Ευρώπη. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στου συμπολίτε μα ότι στην Ευρώπη εφ' δεν υπάρχουν χρήματα για να υλοποιήσουμε τι ε, πολιτικέ ρύθμιση. Ε, αν ε, δεν υπήρχε το Κοινοβούλιο, θα είχαμε πάρα πολύ χαμηλό προπολογισμό για την ΕΣΜΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών κτλ. Δεν μπορούμε δηλαδή να ζητούμε χρήματα και τελικά να μην δίνουμε σε αυτού στους οργανισμούς ε, τα μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους ε, και αν ε, τα μέλη αυτού του κοινοβουλίου δεν μπορούν να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες παρά μόνο στα αγγλικά θα σκοτώσουμε την Ευρώπη. Πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες σήμερα είναι να μπορεί η Ευρώπη να κάνει τη δουλειά της και πραγματικά Εκπλήσουμε που να λένε κάποιοι ότι δεν είναι χρεωμένη η Ευρώπη και μπορεί να δανειστεί και δεν μπορούν να δανειστούν τα κράτη πλέον αλλά η Ευρώπη μπορεί να δανειστεί για να, για να επενδύσει. Ε, αλλά κοιτάξτε, για να μπορεί κάποιο να δανειστεί πρέπει να έχει και ένα προπολογισμό που να το επιτρέπει να αποπληρώσει τα χρέη. Και σήμερα δεν είμαστε στην κατάσταση αυτή. Δηλαδή, εδώ τι λέμε αστεία, να λέμε ότι έχουμε ένα προπολογισμό λιτότητα, ότι μπορούμε να τον ε, διαχειριστούμε ε, με στενότητα. Ε, ε, αυτό εντάξει, αλλά α μην κάνουμε του ανθρώπου να πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρχει προπολογισμό θα υπάρχει μέλλον για την Ευρώπη. Και αν κάνουμε καμερικοπέ, α κάνουμε περικοπές σε άχρηστα πράγματα. Έχουμε τόσα ταξίδια, τόσες αποστολές που είναι άχρηστα. Έχουμε πάρα πολλές δαπάνες για να αγοράσουμε gadget. Να, οικονομίες που μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι τεράστιες, αλλά αν κάνουμε ε, οικονομία κάπου εδώ και εκεί, τελικά πράγματι θα κάνουμε οικονομία. Και ε, φανταστείτε στην δική μου κοινότητα με 300 ε, κατοίκους μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Αν μετρούσα προχωρούσαμε σιγά σιγά, ίσω ε, θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα του λογαριασμού και δεν θα είχαμε τα προβλήματα που περιγράφετε. Σα ευχαριστώ. Thank <clears throat> ε, Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Με σαφήνεια υπέρ μια ισορροπία είμαστε να εξοικονομήσουμε κονδύλια εκεί που μπορούμε, αλλά και με εποπτεία σωστή μια σειρά αποφάσεων μπορούν να εφαρμοστούν και είναι αυτές οι βασικές αρχές να θεσπίσουμε προτεραιότητες υπό το πρίσμα της Οικονομικής και Νομιματικής Επιτροπής πρέπει να συνεχίσουμε με, τα δημοσιονομικά θέματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Πρέπει να έχουμε επαρκή κονδύλια στην Ευρώπη για να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά με το σωστό τρόπο. Στην ουσία είναι θέμα δημοκρατίας αυτό το πρόβλημα ποιο είναι. Απαιτεί λήψη μέτρων το πρόβλημα. Και επιπλέον συνεχίζουμε κάθε μήνα να προσπαθούμε με νέα νομοθεσία να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να ικανοποιήσουμε μια ολόκληρη σειρά νέων απαιτήσεων όσον αφορά τις εξελίξεις. Και ο προπολισμός πρέπει να διευρύνεται με τον ίδιο ρυθμό με τον οποίο διευρύνονται αυτά τα καθήκοντα. Είμαστε υπεύθυνοι για μια σειρά θεμάτων που δεν μπορούν να υποβαθμιστούν. Πρέπει λοιπόν να θεσπιστούν αυτές οι προτεραιότητες ώστε να είναι σεβαστές από τους εμπλεκόμενους ε, ε, απέναντι σε αυτούς που εμπλέκονται στην αγορά για να υπάρξει σταθερότητα στις αγορές και στην οικονομική νομισματική δράση. Χρειαζόμαστε υποστήριξη σε αυτό το, έργο και στην, ε, ε, στο ΕΚΟΦΗΝ θα πρέπει να δοθούν τα αναγκαία κονδύλια και το, και το δυναμικό για να υπάρξουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Σε αυτά τα σχέδια και προγράμματα πρέπει να ζητήσουμε το six-pack, το b-pack που θα αρχίσουν να ισχύουν από του χρόνου και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κιόλας και από το φθινόπωρο. Μια ολόκληρη σειρά χρονοδιαγραμμάτων υπάρχουν, όλο και πιο απαιτητικά χρονοδιαγραμμάτα και στην Ευρω... στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά απαιτούν να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτό το έργο και να έχει επαρκή κονδύλια για να λειτουργήσουν όλα αυτά σωστά. Επιπλέον υπάρχουν δύο και ίδιες κυριότερες προτεραιότητες που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Βελτίωση των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων. Είναι ένα πρόγραμμα αυτό που πρέπει να βελτιώσει τα θέματα τα δημοσιονομικά μέσω αυτών των δράσεων. Σε τοπικό επίπεδο τώρα και σε, και σε σχέση με τα διάφορα όργανα πρέπει να βελτιώσουμε τα μέτρα όσον αφορά τα διαθέσιμα κονδύλια. Στην δημοσιονομική συνεργασία έχουμε ένα μεγάλο δυναμικό που διανοίγεται μπροστά μας ώστε να μπορέσουμε να σταθμίσουμε και να δώσουμε σωστή δράση και να δώσουμε ανακούφιση σε κράτη τα οποία περνούν μέσα από κρίση. Εγώ από πλευράς μου είμαι υπέρ αυτής της ε, επικοδομητικής και ενδιαφέρουσας προσέγγισης. Ελπίζω, ευελπιστώ ότι θα βρούμε λύσεις ώστε να μπορέσουμε να επομιστούμε τις ευθύνες μας, διότι έχουμε μια ολόκληρη σειρά νέων αρχών και οργάνων και λόγω της κρίσης χρειαζόμαστε αυτές τις αρχές και τα όργανα εποπτείας. Όλοι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά σε αυτό το εγχείρημα σε αυτό το εγχείρημα ελέγχου και εποπτείας. Και αυτά τα όργανα χρειάζονται κονδύλια για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλά. Γιατί διαφορετικά γιατί τα θεσπίσαμε και τα δημιουργήσαμε. Ευχαριστώ εσείς για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λαβία μας περιγράψε πολύ καλά το πώς λειτουργεί ο προπολογισμός της Ένωσης στην περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Είμαστε στο τελευταίο τμήμα της ε, επταετούς ε, προγραμματικής περίοδου. Αυξάνονται οι πληρωμές και έχουμε προβλήματα γιατί οι Υπουργοί Οικονομικών δεν καταλαβαίνουν το σύστημα που δημιούργησαν οι ίδιοι και δεν θέλω να πληρώσουν τους λογαριασμούς που δημιούργησαν. Συγκεκριμένα για τον προϋπολογισμό αρμοδιότητας της Επιτροπής μας συμφωνώ με τους κυρίους Γκοζές και Λούδβιξον και οπωσδήποτε πρέπει οι εποπτικές αρχές να έχουν τα κονδύλια που χρειάζονται για να κάνουν την δουλειά τους και έχουν όλο και περισσότερη δουλειά. Και πρέπει να πω πως εάν εντός του προπολογισμού της Επιτροπής μας εξοικονομήσουμε κάτι, θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Γιατί έχουμε μικρό άμεσο κομμάτι του προπολογισμού και από όσο θυμάμαι, πέρα από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ε, είναι κάτι μικρές επιδοτήσεις ε, στην ΣΕΠΣ και κάτι τέτοιες οργανώσεις τότε είναι σε ιδιαίτερη κατάσταση η Επιτροπή μας. Είναι πολύ δύσκολο εμάς να βρούμε κάτι να εξοικονομήσουμε. Και κατά κανόνα όταν το Κοινοβούλιο συζητά τον προπολογισμό εξετάζουμε όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίε από όλες τις επιτροπές γιατί χρειαζόμαστε βεβαίω οι υπηρεσίε αυτές οι ρυθμιστικές να λειτουργούν. Και ο κύριος Φόξ πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Εκτός αν είναι μάγος. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να βρει τρόπο να κάνει οικονομία. Επίσης, να επικρατήσει όταν σα είπε ο κύριος για τον προπολογισμό της Κομισιόν. Πρέπει να μπορούν να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντά τους. Η Κομισιόν βλέπουμε προσπαθεί να ανταποκριθεί στην δέσμευσή της που λέει θα κόψουμε τη διοίκηση κατά 5% και έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε κάποιους τομείς πρέπει να αυξήσουν, σε άλλους να μειώσουν. Είναι καλό αυτό βεβαίως, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και να προσέξουμε μην καταλήξουν να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να μπορούν να έχουν αποτελέσματα στα στατιστικά στοιχεία, στους ελέγχους. Ευχαριστώ Σβέν. Α, όλε. Σε ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να εγκαταλείψω την αίθουσα και δεν θα μπορέσω να ολοκληρώσω και να παρακολουθήσω, να παρακολουθήσω τη συζήτηση πλήρω. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά πρέπει να φύγω για να πάω να ψηφίσω σε άλλη επιτροπή. Αλλού. Ευχαριστώ. Okay. Well, thanks for... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την ε, ανταλλαγή, την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για αυτό το θέμα του προϋπολογισμού για τα δημοσιονομικά. Εμείς ως Οικονομική Νομισματική Επιτροπή έχουμε περιορισμένες, πολύ περιορισμένες ευθύνες. Δεν είναι μεγάλο το τμήμα του προϋπολογισμού που έχουμε ευθύνες. Οι μεγάλες αντιπαραθέσεις για το μέγεθος των δαπανών, για το μίσο που δεν επαρκούν οι δαπάνες, αυτές δεν είναι θέματα ε, του προπολογισμού της ε, ΕΚΟΝ. Είναι λοιπόν μεγάλα θέματα πώς δαπανάει η Ευρώπη τα κονδύλια. Δαπανούμε πολλά κονδύλια σε μία ή πολιτικές. Συμφωνώ με κάποια πράγματα από αυτά που αναφέρθηκαν. Δαπανούμε για μέσα και τρόπους παραγωγής που δεν είναι συνεπείς και δεν συνάδουν με περιβαλλοντικές ε, πτυχές και στόχους στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Αν δούμε τον τομέα για τη γεωργία στον προϋπολογισμό πρέπει πολλές αλλαγές να γίνουν σίγουρα. Το ίδιο ισχύει για την έρευνα. Το ίδιο και όσον αφορά τμήματα της διαθωτικής, των διαθωτικών πολιτικών. Το γνωρίζουμε αυτό. Αυτά δεν είναι όμως τα κυριότερα θέματα τώρα για τη δική μας αρμοδιότητα. Αν υπάρχει μια προσέγγιση ως ΕΚΟΝ, είναι το να δούμε πώς οι δαπάνες στους άλλους τομείς μπορούν να διαμορφώνονται αποτελεσματικά υπό το πρίσμα οικονομικών πολιτικών. Αυτό ακριβώς θα είναι μια αξιόλογη συζήτηση σε σχέση με τα θέματα του εισηγητή. Και θα είναι μια αξιόλογη συζήτηση επί της ουσίας, λέω. Αξιόλογη συζήτηση επαναλαμβάνω. Πέρα από όλα αυτά, ο ε, τα θέματα προϋπολογισμού από πλευρά ΕΚΟΝ δεν είναι ε, το σημείο για να δώσουμε τις αντιπαραθέσεις υπέρ ή κατά κυβερνητικών δαπανών ή δαπανών από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση έστω. Ε, οι διάφοροι οργανισμοί και υπηρεσίες φορείς, το έχουμε συζητήσει ανοιχτά, επανειλημμένα για την υλοποίηση και ενίσχυσή τους μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, ιδιαίτερα που ε, είχαμε εμεί ιδιαίτερα οι υποπτικές ε, ε, υπηρεσίες και όργανα είναι, όργανα. είναι καλή θετική επένδυση για την Ευρώπη. Αν ήταν δυνατόν με περισσότερε εξουσίε και νωρίτερα να έχουν γίνει κάποια πράγματα, θα είχαμε εξοικονομήσει δαπάνε και κόστη. Είναι ηρωνικό να ζητά κανεί τώρα να υπάρξει μείωση των κονδυλίων για τι ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ, όταν προέρχεται αυτό από μια χώρα που έχει τόσο πληγεί αρνητικά όσον αφορά την αρνητική εποπτεία και δεν πρέπει να επαναλάβουμε τέτοιου είδους σφάλματα. Πέρα από όλα αυτά, η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει επανειλημμένα ζητήσει και έχει πει ότι οι οργανισμοί αυτοί και οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν επαρκή κονδύλια και όρους εργασίας για να υλοποιήσουν τους στόχους και το έργο που ε, ε, επομίζονται μέσω νομοθεσίας. Πρέπει να είμαστε ε, συνεπείς σε δύο επίπεδα. Δεν μπορούμε νομοθετικά όλο και περισσότερες αρμοδιότητες να μεταθέτουμε στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και μετά στη συνέχεια να, τους, να στερούμε από αυτές τα αναγκαία κονδύλια και το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό στη στελέχωσή του. Πρέπει να είμαστε συνεπεί και συνεκτικοί λοιπόν εδώ. Και δεύτερον, πρέπει να είμαστε συνεπεί και συνεκτικοί όσον αφορά επίση την το μέγεθος, το εύρος του προϋπολογισμού. Σε βάθος εργαστήκαμε όσον αφορά το πλαίσιο της Επιτροπής Αντιμετώπισης της Κρίσης. Ο Βόλφ Κλίνς ήταν ο πρόεδρος εκεί. Έχουμε ισχυρέ θέσει ω Ευρωβουλή για τα θέματα τα δημοσιονομικά σε αυτή την πτυχή. Να μην ξεχνάμε λοιπόν αυτά που έχουμε ήδη συμφωνήσει στο παρελθόν. Και θέλω να έχουμε καλή συνεργασία σε σχέση με τις θέσεις ε, από πλευρά εισηγητού. Να μην τεθούν οι, δικές, οι προσωπικές απόψεις στο επίκεντρο, αλλά οι αποφάσεις της δικής μας Επιτροπής και της Ευρωβουλής ευρύτερα. Ευχαριστώ. Ε, ναι, ευχαριστώ. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Πρώτα απ' όλα υποθέτω πως κάθε δημόσιος προϋπολογισμός είναι υποχρεωμένο, υποχρεωμένος από τον νόμο να είναι ισορροπημένος ε, ε, και υποθέτω πως αυτό συμβαίνει. Και τα έξοδα, αν δει κανείς, αν θέλει να ασκήσει κριτική στα έξοδα της γεωρικής πολιτικής, εντάξει, μπορεί, αλλά υπάρχει και πολιτική αιτία. Είναι η διατροφική ασφάλεια που έπρεπε να διασφαλιστεί μετά τους παγκοσμίους πολέμους στην Ευρώπη. Βεβαίω σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική, αλλά δεν είναι. νομίζω πως μπορεί να γίνουν πράγματα με τρόπο αυθαίρετο. Να υπενθυμίσω πως ε, συνολικά δε, ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό είναι 1% του ΑΕΠ της ε, κοινότητας. Ε, είναι μεγάλο ποσό, αλλά δεν είναι συνολικά μεγάλο ποσό συγκρινόμενος με το ΑΕΠ τη κοινότητα και νομίζω πως σε γενικές γραμμές χρησιμοποιείται λογικά. Έχουμε επίσης μπροστά μας διευρύνσεις. Θα ενταχθεί και η Κροατία και θα έχουμε βεβαίως ανάγκες για νέες αγροτικές πληρωμές και περιφερειακά κονδύλια. Το 2004 είχαμε μια τεράστια διεύρυνση, πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Και έχουν ανέβει κατά πολύ περισσότερο οι προπολογισμοί των κρατών μελών από, τις, ε, από ό,τι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε νομίζω πως μπορούμε να πούμε πως χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά. Εγώ θα ήμουν ακόμη πιο επιθετικός. Θα έλεγα πως αυτή τη στιγμή χρειάζονται περισσότερα λεφτά δεδομένων των ε, ε, περισσότερων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκή Ένωση Για τι δε υποπτικέ αρχές ακούσαμε κάποια πράγματα και εγώ συμφωνώ. Δεν είναι κόστος οι αρχές αυτές, είναι επένδυση. Και στόχο έχουμε βεβαίως να αποφύγουμε κρίσεις. Ναι. Αυτά είχα να πω δεν θα μιλήσω περισσότερο. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε στην Επιτροπή μας για μια σταθεροποίηση του προπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε περάσει τώρα στο χρόνο του επόμενου θέματος και έχουμε ακόμα τρία, τρεις συναδέλφους να μιλήσουν. Βίκη, ευχαριστώ. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη που ξεκινά νωρίτερα αυτή η διαδικασία στο δημοσιονομικό έτος, γιατί στο παρελθόν ε, τα, κατά κάποιο τρόπο συζητήταν αυτό ε, στο Φερινό, στις θερινές διακοπές και αυτή η Επιτροπή δεν μπορούσε να δράσει με τη δέωση επιμέλεια, δηλαδή να συζητήσει με τους αρμόδιους για τη δαπάνη των γραμμών προπολογισμού και νομίζω ότι Τώρα η διαδικασία αυτή μας βοηθά να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ε, και ανεξάρτητα με το αν υπάρχουν πιο ξυπνοί τρόποι να συνεργαστούμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο με τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών. Ε, νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να δούμε ποιες γραμμές προπολογισμού δεν έχουν δαπανηθεί ε, παρκώς στον προπολογισμό και μπορούν να μειωθούν, να έχουμε περικοπές και να δούμε πιο μακριά πέρα από το ένα έτος στην οδηγία για τη δημοσιονομική οικονομικό πλαίσιο ζητήσαμε από του ηγητέ να δουν τον αντίκτυπο στον προπολογισμό και νομίζω ότι μπορεί να δώσει το παράδειγμα αυτή η Επιτροπή όχι μόνο να εξετάσει τι δικέ τη γραμμέ προπολογισμού σε πρόθεσμα αλλά ίσω να κάνουμε και κάποια γενικά σχόλια για τι γραμμέ προπολογισμού αλλού και πάλι στο παρελθόν είχαμε διάφορα θέματα για τα συνταξιοδοτικά συστήματα ε, και για το αν συνάδουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τον κρατών μελών. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον συγγητή για το έργο του. Ευχαριστήσω τον συγγητή πρώτα απ' όλα. Τώρα για τις ε, γραμμές εκείνες δαπανών που δεν εξαντλώνται γιατί δεν είναι σε θέση παραδείγματο χάρη στα διαρθρωτικά ταμεία να απορροφήσουν ε, τα κράτη-μέλη, τα κονδύλια αυτά τα οποία υπάρχουν στον προπολογισμό και η Κομισιόν ε, συχνά επικρίνεται για το ότι δεν θέλει να διαθέσει αυτά τα κονδύλια ενώ δεν είναι σε θέση να αλλάξει την κατανομή. Γι' αυτό το ερώτημά μου προς τον συγητή είναι είναι διατεθειμένος η πολιτική αυτή να αλλάξει, δηλαδή να μπαίνουν τα κονδύλια αυτά στα διαρθρωτικά ταμεία και να υπάρχει δυνατότητα μετά να πάνε αλλού για να χρησιμοποιηθούν ε, αποτελεσματικότερα και να χρησιμοποιηθούν τελεία. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που είναι εναντίον, αλλά νομίζω πως θα πρέπει να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και τελευταίος μιλητής είμαι εγώ η ίδια. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στη τελευταία ολομέλεια για την έκθεση προπολογισμού ψηφίσαμε μια τροπολογία που έλεγε ότι το είναι προτεραιότητα και έπρεπε επίσης ε, να υπάρχει παροχή ανεξάρτητων νομικών συμβουλών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα καθώς ε, προχωρούμε γιατί έχουμε ένα μεγάλο αριθμό κατεξουσιοδότηση πράξεων και έχουμε πάρα πολλέ σημαντικά νομικά θέματα. Υποστηρίζω λοιπόν όσο είπαν οι υπόλοιποι για το θέμα ότι πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα για τους οργανισμούς αυτούς για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρούμε αυτό σε ένα προϋπολογισμό σχεδόν de που έχουμε εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να δούμε τι υπόλοιπε υπηρεσίε, του υπόλοιπου οργανισμού και να πούμε να μην αυξήσουμε συνολικά τι δαπάνε για του οργανισμού ή να εφαρμοστεί κάποιο άλλο μέσο, κάποιο άλλο εργαλείο, γιατί συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν προπολογισμό που θα ακολουθεί τον πληθωρισμό. Όμω ε, πολλοί ταυτόχρονα ε, δεν θέλουν να κόψουν τον προπολογισμό αυτών των οργανισμών και τι δημοσιονομική σταθερότητα και ξέρετε ότι και αυτό είναι ένα από του λόγου που είμαστε σε αυτή τη λιτότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ λοιπόν κυρία Λαβία. Ήδη τρώμε χρόνο από το επόμενο θέμα, τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει και την δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά θέλετε το λόγο για δύο λεπτά, θα σα τον δώσω. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και αυτό είναι ο πραγματικός λόγος που ζητάει ο συγγητή ε, ακρόαση από τις ειδικέ επιτροπές, γιατί ακριβώς ε, ζητάμε να συλλέξουμε ειδικά στοιχεία σε σχέση με τις προτεραιότητε των διάφορων επιτροπών. Η δική σα ε, συνεισφορά είναι προφανής και ήδη είχε προταθεί στις κατευθυντηρίες γραμμές ε, ότι δεν ήταν ε, ο κατάλληλος τόπος να ε, τοποθετηθεί το θέμα των προτεραιοτήτων αλλά στον, στην εντολή του τριμερούς διαλόγου θα βάλουμε τις προτεραιότητες που θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως το θέμα είναι πολύ σημαντικό είναι ζωτική σημασία. Ε, πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε μόνο να ζητάμε. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που θα στείλουμε. Δεν μπορούμε να ζητάμε περισσότερα. Μόνο θα πρέπει και στο πλαίσιο του συνολικού προπολογισμού να εντοπίσουμε κάποια προγράμματα τα οποία έχουν χαμηλά επίπεδα εφαρμογής ή προγράμματα που δεν ε, είναι ύψης της σημασίας στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων μας για να γίνει κάποια αναθεώρηση Έγινε μία σειρά παρατηρήσεων, είναι σαφές ότι οι δικές σας ε, προτεραιότητες θα τις καθορίσετε εσείς ε, στη δική σας επιτροπή. Εγώ, αφού σας άκουσα όμως μετά από αυτό τον πρώτο γύρο τραπέζης, ε, στον τριμερή διάλογο θα συμπεριλάβω αυτά τα στοιχεία και φυσικά οι τραπεζικέ αρχέ πρέπει να έχουν του απαραίτητους φόρους για να λειτουργήσουν σωστά. Κατόπιν έγινε συγκεκριμένε ερωτήσει σε σχέση με τι περιφερειακές πολιτικέ, αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι αυτέ οι πολιτικέ έχουν μία προσέγγιση προ τα κάτω. Έτσι λοιπόν ο επαναπρογραμματισμό θα γίνει από τα κράτη-μέλη, από τι ενδιαφερόμενε περιφέρειες. Είναι σαφές ότι στο πλαίσιο ε, των κονδυλίων που διατίθεται, ο καθένα πρέπει να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του ε, πόρου που διαθέτει. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Και έτσι λοιπόν ε, πρέπει να ε, μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους αυτούς με τον κατάλληλο τρόπο στις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θα εξετάσουμε το σχέδιο της ε, γνωμοδότησης ε, στις 30 Μαΐου ή στις 19 ε, Ιουνίου, πιθανόν. Και αν είναι δεύτερη ημερομηνία δεν έχει νόημα. Η ημερομηνία που έχω εδώ για την προθεσμία κατάσταση προπολογισμών 18 Ιουνίου, αλλά θα εξετάσουμε τροπολογίες στις 10 Ιουλίου και θα ψηφίσει η Επιτροπή Προπολογισμού τον Οκτώβριο, αλλά το επόμενο θέμα θα είναι λοιπόν το σχέδιο τη γνωμοδότηση. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, σημεία 8 και 9. Έχουμε την οδηγία και τον κανονισμό για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει και θα έχουμε μία ανταλλαγή απόψεων επί των τροπολογιών. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Τμαρκάρας. Πρόεδρε, σας χαιρετίζω στο διπλό ρόλο σας ως κοιόδους εισηγήτρια της ομάδας και ως πρόεδρο για αυτό το χαρτοφυλάκιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, εισαγωγικά θα ήθελα τέσσερα σημεία να θέσω υποσυζήτηση και να παρατηρήσω επ' αυτών κάποια πράγματα. 1643 τροπολογίες κατατέθηκαν για αυτόν τον κανονισμό. 552 τροπολογίες όσον αφορά την οδηγία την ίδια. 2.195 λοιπόν συνολικά τροπολογίες. Λοιπόν, για μένα ως εισηγητή θετικό είναι βέβαια και διευκολύνει το έργο μου το γεγονός ότι όλες, σχεδόν όλες οι τροπολογίες στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Πράγμα το οποίο φυσικά οφείλεται τελικά στο ότι είχαμε μια σε βάθος συζήτηση κατά τη διάρκεια του 2010 και στη συνέχεια μετά για αυτά τα θέματα από το 2010 και μέχρι σήμερα. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπλέκεται και συντάσσεται έτσι μέσα στους στόχους αυτούς που εμείς διατυπώσαμε ως Ευρωβουλή. Δεύτερη παρατήρηση. Εργαζόμαστε με πλήρη ρυθμό για συμβιβασμούς και θέλω σε σχέση με τους συνεργάτες της Επιτροπής μας και τους συνεργάτες των Ευρωβουλευτών να ευχαριστήσω για αυτό το έργο. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και όσον αφορά χρόνο και όσον αφορά το αποτέλεσμα ήταν αναγκαίο και καταφέραμε να πετύχουμε θετικά πράγματα. Όλοι λένε λόγω του μεγάλου αριθμού των τροπολογιών και λόγω των δυσκολιών που συναρτώνται με αυτό το θέμα ότι είναι αναγκαίο τώρα να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα και να το προσαρμόσουμε Παρακαλώ να μην κάνουμε κάτι τέτοιο, να απόσχουμε από κάτι τέτοιο στόχο. Είναι φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, είναι φυκτό, μπορεί να τηρηθεί και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πω ότι πρέπει, θα ήθελα να το τηρήσουμε και προς όφελος εκείνων που εμπλέκονται στις αγορές και για ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μέσα στο πλαίσιο της ε, διατύπωσης της κοινής θέσης, ε, επίτευξης κοινής θέσης του Συμβουλίου. Ελπίζω ότι θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και στις 25-26 Απριλίου στο τέλος τέλος στην Οικονομική Νομισματική Επιτροπή θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε προς έγκριση. Τρίτον, αναμένουμε ακόμα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για παράδειγμα την έκθεση από πλευράς της που ζητήσαμε να συνταχθεί όσον αφορά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί και σημειώνται στην διαδικασία ε, της Βασιλείας και και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά. Τέταρτον, στις τροπολογίες ε, υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις σε σχέση με την δική μας σχέση ε, για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις από συντάκτες τροπολογιών ότι υπάρχει δυσανάλογη ίσως ε, τοποθέτηση έναντι του ΕΠΕΡ και θα μπορούσαν τα μικρότερα όργανα ή ε, οργανισμοί να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις. Κατανοώ αυτές τις επιφυλάξεις. Θα ήθελα να πω στα μέλη της Επιτροπής ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά όσον αφορά αυτή τη διαδικασία του ΕΠΕΡ και θα είμαστε κάθε στιγμή έτοιμη να ε, υπάρξει ενημέρωση και να υπάρξει εξέταση των προτεραιοτήτων και χρονοδιαγραμμάτων έγκαιρα. Όλοι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε, επιτρέψουμε ότι από, μια, ε, από ένα οργανισμό θα πρέπει να γίνεται πολιτική. Πολιτική πρέπει να γίνεται από εμάς που είμαστε οι Και σε συνεργασία με το θα πρέπει εκείνες οι αποφάσεις να μπορούν να ληφθούν, αποφάσεις από πλευράς μας ε, που ας το πω έτσι κλιμακώνονται, μπορούν έτσι αλληλοδιάδοχα να επενεργούν όσον αφορά τις προτάσεις μας. Ταυτόχρονα υπάρχουν όμως όσον αφορά και τις τροπολογίες πάρα πολλές που περισσότερο από πλευρά της αποσαφήνισης ε, αφορούν την πτυχή ΕΠΕΡ και πρέπει αυτές να τις συζητήσουμε σίγουρα. Ο ίδιος, προτού περιστραφώ και εξετάσουμε τα επιμέρους κεφάλαια, παρακαλώ να λάβουμε υπόψη σε τρεις τομείς τα θέματα των τροπολογιών που πρέπει να εξεταστούν υπό το φως συζητήσεων που έχουν ήδη γίνει με τους συναδέρφους. Μία τροπολογία αφορά τη μείωση των κινδύνων όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τονίζω όμως εδώ ταυτόχρονα μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι για το συνολικό χαρτοφυλάκιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, θέλουμε να στηρίξουμε και να ε, ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις μας. Όμως πρέπει να, να, είμαστε, ε, να λαμβάνουμε υπόψη την αναλογικότητα. Και όσον αφορά κατόφλια και κάποιες τροπολογίες ε, που προτείνουν τέτοιου είδους κατόφλια, μετά από αίτημα της Ευρωβουλής και σε ε, σύντονη δράση της ε, Επιτροπής ε, εξετάζεται η τροποποίηση, η προσαρμογή σε σχέση με τα κατόφλια, με τις τιμές αυτές και αναμένουμε το αποτέλεσμα. Επιπλέον έχουμε και συστημικά σημαντικά όργανα που μπορούν να ληφθούν υπόψη και σε σχέση με την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου που μπορεί να οδηγήσει σε κλειδονισμούς πρέπει να βοηθήσουμε με κεφαλαιακές απαιτήσεις να μην υπάρχουν υπερβολικά μεγάλοι κίνδυνοι και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Μόνο σε κάποιες λίγες λεπτομέρειες θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες παρέκκλησης. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Η τρίτη ομάδα τροπολογιών και που από πλευράς ε, εισηγητού ε, προτάθηκε είναι το θέμα της ε, μισθολογικής πολιτικής ή της πολιτικής αμοιβών των τραπεζών corporate governance θα πρέπει από πλευράς ε, ε, να καθοριστούν οι κίνδυνοι και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ταυτοποιηθούν, να εντοπιστούν σε σχέση με συνεργάτες χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος και που πρέπει να δεσμεύονται όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Μέχρι σήμερα ο εντοπισμός, η ταύτιση αυτή γινόταν με αυτοαξιολόγηση των ε, ε, ιδρυμάτων αυτών. Πρέπει να αποφεύγεται όμως ο υψηλός κίνδυνος, το δυσανάλογος κίνδυνος καθώς επίσης ε, και ο καθορισμός των κειμενόμενων αμοιβών. Η προσέγγιση μου είναι δεν πρέπει να είναι η, δια, η κειμενόμενη ε, αμοιβή περισσότερο από το διπλάσιο της ε, κανονικής, του κανονικού μισθού, των κανονικών απολαβών. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτή τη συζήτηση, να κάνουμε το αναγκαίο μόνο, να μην κάνουμε εκείνα τα οποία ε, θα μπορούσε να χαρακτηριστούν, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως λαϊκιστικά. Και όταν έχουμε υψηλά προσοντούχους που εμπλέκονται θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιτελούν υπεύθυνα το έργο τους Τώρα, για το τελευταίο τμήμα, οι τομείς εκείνοι όπου έχουμε τροπολογίες που ε, κατατίθενται και που πρώτον, ο πρώτος τομέας είναι και παραμένει το θέμα του προσδιορισμού του κεφαλαίου, των κεφαλαίων. Πολλές τροπολογίες υπάρχουν για τον ορισμό των διαφορετικών κεφαλαιακών μέσων κεφαλουχικών μέσων. Εγώ πιστεύω ότι με σαφήνεια πρέπει να τοποθετηθούμε και να πούμε έχουμε μια προσέγγιση επί της ουσίας substance of form approach. Τώρα πρέπει όμως να εξειδικεύσουμε τα, τις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να υπονομεύσουμε τις κεφαλαϊκές απαιτήσει, γιατί τότε θα αποδυναμώσουμε γενικά τη δική μας προσέγγιση όλες οι τράπεζες να αποτελούν ε, αντικείμενο αυτών των, αυτού του κανονισμού και των, της οδηγίας και να λαμβάνονται υπόψη οι μορφές και οι ανάγκες τους. Για τις ε, πιστώσεις ε, προσεγγίζουμε με ενιαίο τρόπο το πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι πιστώσεις αυτές και η έγκρισή τους. Κάποιοι ευρωβουλευτές έχουν σε ποσοστό την ε, μείωση που προβλέπεται. Άλλοι σε κλιμακούμενη, σε κλίμακα που προτείνεται. Θα πρέπει εδώ να δούμε και το θέμα των ορίων ηλικιακών και άλλων. Όλες αυτές οι προτάσεις ε, εντάσσονται στο πλαίσιο αυτό και το θέμα της ε, μείωσης του ποσοστού κατά ένα τρίτο καθώς επίσης και το θέμα της αύξησης του ορίου η στάθμιση ε, κρατικών ε, δανείων και πιστώσεων και αυτή είναι ε, σημαντική υπόθεση. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι ευρωβουλευτές να, λαμβάνουν, να λαμβάνεται υπόψη το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Άλλοι να αναμείνουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και μετά να έχουμε παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, χρειαζόμαστε μια νέα στάθμιση κινδύνων όσον αφορά τα κρατικά δάνεια, τα δημόσια δάνεια. Όμως οι συνέπειες μέσα από τη διαδικασία της Βασιλείας έχει σίγουρα δημοσιονομικές και νομισματικές επιπτώσεις. Στο δεύτερο τομέα, εδώ θα πρέπει σε σχέση με την ρευστότητα να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Τίθεται το ερώτημα αν η αναλογία ρευστότητας είναι επαρκής ή αν θέλουμε νωρίτερα να εφαρμοστεί. Το ίδιο όσον αφορά την αναλογία για την ε, ε, εξέλιξη του προγράμματος χρονικά. Και εδώ πάλι δεν θέλω να υπάρξουν καθυστερήσεις σε σχέση με αυτά τα μέτρα. Αν εντοπίσαμε και αναγνωρίσαμε σε σχέση με την έκθεση πρωτοβουλίας ότι είναι αναγκαία αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό θέλουμε να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στο θέμα της ρευστότητα. Το εντάξαμε στις ε, εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να αναμείνουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε όλα τα εργαλεία, τα μέσα στο τραπέζι για να δούμε τι πρέπει να γίνει για τη ρευστότητα. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πλευράς ΕΠ λοιπόν μπορούμε να ζητήσουμε να γίνουν όλα αυτά αποτελεσματικά. Μόνο έτσι θα ε, διασφαλίσουμε ώστε να μπορούν οι πληρωμές έγκαιρα να ε, διεξάγονται και να ενισχυθούν έτσι να ενδυναμωθούν οι τράπεζες. Τρίτο, τρίτη κατηγορία, αναλογία μόχλευσης, ε, ποσοστό μόχλευσης. Θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αν στον πυλώνα 1 ή πυλώνα 2 θα πρέπει να ενταχθεί ως μέτρο. Ως μέτρο πυλώνα ένα θα έπρεπε να διαφοροποιήσουμε τα πρότυπα της, ε, του επιχειρηματικού προτύπου ε, είναι νομίζω κάτι το γνωστό αυτό και πορεύονται προς αυτήν την κατεύθυνση αρκετοί ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτό με συνεκτικό τρόπο να το εντάξουμε. Η περίοδος αξιολόγησης θα πρέπει λοιπόν να λειτουργήσει και να αναμείνουμε να ολοκληρωθεί και να δούμε τα αποτελέσματα. Τελευταίο θέμα η λειτουργικότητα ή η δράση σε σχέση με ελάχιστο επίπεδο ή μέγιστο επίπεδο. Χρειαζόμαστε σίγουρα την ελαστικότητα, την ευελιξία. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και θα έχει ε, μια εποπτική δραστηριότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δράση Διαφάνεια και κοινοί κανόνες λοιπόν απαιτούνται και συντονισμός όλων αυτών μέσα από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό στον κανονισμό σε σχέση με την πρόταση όσον αφορά κάποιο κράτος μέλος που υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ε, μετά από έγκριση και εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ξεπεράσει κάποια συγκεκριμένα όρια. Θα πρέπει να ε, επεξηγεί αυτό το συγκεκριμένο κράτος μέλος ποιοι κίνδυνοι ε, αναγκάζουν αυτή την παρέκκληση και θα πρέπει να δούμε και την υποχρέωση δημοσιοποίησης υπό το αντίστοιχο άρθρο από, σε σχέση με το 418 ή 440 που θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε και την πρόταση για το ίδιο κεφάλαιο από κοινού με την ε, ε, γενικότερη προσέγγιση δίνει επαρκή ελαστικότητα όσον αφορά τις κεφαλαϊκές ανάγκες. Σε σχέση με το άρθρο 443, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υιοθετεί συγκεκριμένα μέτρα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό το διευρύνουμε εμείς. Στο τέλος θα ήθελα να πω και να ολοκληρώσω ότι και ο κανονισμός και η οδηγία θα πρέπει για όλους να ισχύουν. Έχουμε πληθώρα τροπολογιών που αποκλειστικά αφορούν εθνικές ιδιομορφίες ή ε, στοιχεία ή συγκεκριμένες ανάγκες ε, εθνικά ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτές δεν πρέπει να απεμποληθούν, να αγνοηθούν. Όμως ο κανονισμός ή η οδηγία μπορούν μόνο να λειτουργήσουν σωστά όταν έχουμε ένα level playing field, ένα ισοδίκαιο πλαίσιο λειτουργίας και προσέγγισης για όλους, που θα ισχύει για όλους. Εδώ θα πρέπει να διεξαχθούν επαφές και συζητήσεις. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το θέμα της συνένεσης. Συνένεσης και από πλευράς των πολιτών μας και των κρατών μελών που αποτελούν προϋπόθεση για αυτά τα μέτρα και τη σωστή τους λειτουργία. Στόχος μας ε, και σκοπός μας είναι να υπάρξουν ρυθμίσεις και κανονισμοί για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην αγορά θα πρέπει να σέβονται αυτές τις αρχές. Θα πρέπει η εσωτερική αγορά να διασφαλιστεί και ένα ισοδίκαιο πλαίσιο λειτουργίας ώστε ο χρηματοπιστωτικός τομέας να καλυφθεί επαρκώς. Δεν κάνουμε εξαιρέσεις δεν κάνουμε εξαιρέσεις και σίγουρα δεν θα προτείνουμε να υπάρξουν περαιτέρω εξαιρέσεις ή να εξεταστούν άλλες εξαιρέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, υπό αυτή την προσέγγιση ζητώ να υποστηριχθεί αυτό το έργο. Θα έχουμε αυτή την εβδομάδα μια συνάντηση σκιωδών εισηγητών που θα συναντηθούν, θα υπάρξουν συζητήσεις και επαφές με επιμέρους ευρωβουλευτές, με εμπλεκόμενους στις ε, αγορές. Θα ήθελα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή να μην ε, εμπλακούμε σε αυτό το εγχείρημα με ξένους, με ε, εξωγενείς παράγοντες καλύπτουμε έτσι όλες τις πτυχές. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην εξετάζεται και να μην καλύπτεται μέσα από αυτό το δίκτυο των τροπολογιών. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να υποβάλει λοιπόν την πρόταση προς ψήφιση και έγκριση δεν έχει κανένα, νόμο, κανένα νόημα να εμπλακούν τώρα εξωγενείς παράγοντες και να συζητήσουμε με άλλους ξένους. Εμείς είμαστε αρμόδιοι και μεταξύ μας πρέπει να βρούμε μια βάση συνεννόησης για να υπάρξει συνένεση και να υπάρξει ευρεία υποστήριξη μετά στην ψήφιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ μου έχουν το λόγο και νομίζω ότι πρέπει να έλεγξω τον κατάλογο. Θα το διαβάσω για ανά ομάδες. Δεν θα τα πω με τη σειρά. Νούτα Χουμπνε, Κόριν Βερτμαν Κούλ, Αστρίντ Λούλινγκ, Γκούνα Χόκμαρκ, Άνδρια Σουάμπ, Παμπλο Ζάλμπα, Πίτερ Ζήμον, Άν Γένσεν, Βουλφ Κλίντσεν, Σίλβι Γκούλαρντ. That is in addition to the... Και αυτή είναι πρόσθεση, προσθήκη στους Κιαωδείς. Εγώ, Φόρτ, Φιούτ, ο κύριος Ντόρφαν επίσης ε, μας ζήτησε το λόγο και ο κύριος Νίτερης. Ε, και μπορεί να συνεχίσουμε και στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων τη συζήτηση. Καταρχήν η ε, και ο εκπρόσωπος των Δημοκρατών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτά τα οποία μας είπε για την πάρα πολλή δουλειά που έχει κάνει εδώ και καιρό για το θέμα αυτό. Επειδή πολλοί είναι οι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν, θα ήθελα οι πολλές προτάσεις μας να συνοψιστούν σε δύο ομάδες και να αφαιρθώ μόνο στα σημαντικότερα σημεία. Πρώτα απ' όλα, σκέψη μας είναι όσον αφορά την ε, αναδιαμόρφωση αυτού του τομέα. Σβήνουμε τα σωστά ή ε, τα λάθος. Γιατί νομίζω πως τελικά θα έχουμε κάποιες ε, συνέπειες μη εσκεμμένες και δεν ξέρω αν θα αντιμετωπίσουμε τις αιτίε των προβλημάτων και θα έχουμε καλύτερη ρύθμιση. Η ομάδα μου έχει την άποψη πως ε, καλά θα κάναμε να λάβουμε υπόψη την ε, πολυμορφία του ε, διαφόρων χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και να την ενισχύσουμε, να μην υπάρχει μόνο ένα ενιαίος τύπος ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο θα καταλήξουμε σε τελική ανάλυση. Έχουμε ένα διαρθρωμένο τραπεζικό σύστημα, ε, το οποίο δεν θέλουμε να καταργήσουμε, θέλουμε να ενισχύσουμε. Και το ερώτημα είναι πώς με αυτόν τον ε, κανονισμό θα μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε όσον αφορά τις διατάξεις ε, ιδίων ε, κεφαλαίων ε, νομίζω θα πρέπει να υπάρξει μια κατάταξη ανάλογα με το μέγεθος του ισολογισμού και του κάθε ιδρύματος. Δεν ισχύουν τα ίδια πράγματα για όλες τις τράπεζες, επιχειρηματικές και λιανικής. Ξέρω βεβαίως πως κάποιοι άλλοι συνάδελφοι κάνουν μια διαφορετική κατάταξη ανάλογα με τους διάφορους τύπους ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε αλλά θεωρούμε πως οπωσδήποτε θα πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις ε, ε, περί ιδίων κεφαλαίων αναλόγως με τον κίνδυνο που υπάρχει όσον αφορά δε το ποσοστό χρέωσης πάλι το ίδιο πρόβλημα έχουμε πώς θα μπορέσουμε το ή με τον ίδιο λόγο χρέωσης ε, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές ε, τράπεζες. Εδώ πέρα θα θέλαμε από την Κομισιόν να κάνει κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε στρατηγικά την ε, συμπεριφορά του κινδύνου στην ε, αγορά και πάλι εδώ πέρα κάποιοι συνάδελφοι έχουν προτείνει να υπάρξει μια κατάταξη ανάλογα με τον τύπο τραπέζης και εδώ πέρα είμαστε υπέρ μια συζήτηση να ζητούμε μια λογική λύση για να αναπτύξουμε και να δούμε διαφορετικά το κάθε προφίλ επικινδυνότητας. Τώρα σε τελική ανάλυση το τι κάνουμε στην ε, πραγματική οικονομία. Έχει μεγάλη σημασία το τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γι' αυτό είμαστε υπέρ μιας ε, σαφούς μείωσης ε, της αξιολόγησης του κινδύνου σε αυτόν τον τομέα και θα το συζητήσουμε αυτό με τον εισηγητή και νομίζω πως ο Ότμαρ Κάρας έχει δείξει ακριβώ μεγάλη κατανόηση για αυτή την πτυχή που έχει σχέση με την πραγματική οικονομία και είναι σημαντική για την ανάπτυξη και τις εργασίες. Είμαστε λοιπόν τώρα στο δεύτερο σημείο το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα, δηλαδή το εάν η ρύθμιση είναι αρκετά ακριβής όσον αφορά την διαφοροποίηση των τραπεζών. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο είναι πώς θα έχουμε ασφάλεια σε ολόκληρο το σύστημα. Ναι, πράγματι θεωρούμε λοιπόν πως πρέπει να έχουμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση για να είναι τα κράτη-μέλη σε θέση να ε, αντιμετωπίσουν την ε, ιδιαίτερη κατάσταση που υπάρχει στο καθένα. Εντάξει, θα είναι ενιαία η νομοθεσία, αλλά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να λάβουμε υπόψη το εάν μια χώρα ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο ε, εφαρμογής της νομοθεσίας που χρειάζεται και άρα υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με αυτό ή εάν Μία χώρα έχει πολύ μεγαλύτερο τραπεζικό τομέα από άλλες χώρες. Ο εισηγητής εδώ πέρα προτείνει να υπάρξει ένας βαθμός ελευθερίας ε, στην εφαρμογή σε συνδυασμό με τον ε, κανονισμό αυτών. Λογικό, είμαστε υπέρ. Τώρα τις λεπτομέρειες μπορούμε να τις δούμε, αλλά επί της αρχής μπορούμε να συνοηθούμε σε ένα κοινό πλαίσιο και μετά τις ε, λεπτομέρειες ε, θα τις δούμε. Είναι σημαντικές. Τώρα, κρατικά ομόλογα, τι θα κάνουμε με αυτά. Αυτοί οι οποίοι λένε πως θέλουν αμέσως μια διαφορετική ε, ένα διαφορετικό υπολογισμό για αυτά. Πρέπει να μας εξηγήσουν και τι εννοούν, τι γίνεται και με πιστώσεις των ε, Δήμων που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές σε πάρα πολλές ε, χώρες. Δεν είναι θέμα μόνο ιδεολογικό και να μην ε, λαμβάνουμε υπόψη τις συνέπειες που θα έχουν. Έγινε λοιπόν νομίζω από μας μια έξυπνη πρόταση όπου λέμε πως μακροπρόθεσμα η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση αλλά μακροπρόθεσμα εμείς θεωρούμε τα ευρωομόλογα τόσο σταθερά ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για μια αξιολόγηση πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό το οποίο δεν έχει καταλάβει το CDU και ο Βέρνερ Λάγκεν είναι πως ε, έχουμε μια πάρα πολύ ε, προστατευμένη θέση των γερμανικών ομολόγων ε, και στο άλλο άκρο βεβαίως ε, έχουμε την αντίστοιχη κατάσταση για τα ομόλογα των νοτιών χωρών. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν ωφελεί. Θα πρέπει λοιπόν να συνεισφέρουν τα γερμανικά ομόλογα στην σταθερότητα την κατάσταση. Τέλος πάντων θα μπορέσουμε να έχουμε μια μια αξιολόγηση των ευρωομολόγων με το μηδέν ως βαθμό επικινδυνότητας, αυτό το οποίο είπατε. Τώρα για τους άλλους συναδέλφους, ε, ο κ. Μπεκάς δεν είναι εδώ, αλλά κορεσοποιείται από τον κύριο Λχαντραουή και έχει καταθέσει κάποιες τροπολογίες. Ε, τέλος, για την ασφάλεια συνολικά του συστήματος όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά και αριθμούς της ρευστότητα. Θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε μια γρήγορη εισαγωγή αυτών των τιμών και ορίων γιατί σε τελική ανάλυση το θέμα ήταν ακριβώς το ότι δεν διαχειριστήκαμε σωστά αυτά τα πράγματα και εντός των ε, προθεσμίων και στην Lehman Brothers και σε άλλες ε, περιπτώσεις. Αυτά κατά την απόψή μου είναι τα σημαντικότερα τα οποία θα μας απασχολήσουν τις άλλες ε, τις ερχόμενες εβδομάδες. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα θεωρώ πως πρέπει να κινηθεί ώστε να τον πιο γρήγορα το Κοινοβουλίο αλλά πρόκειται για ένα τόσο τεράστιο και σημαντικό θέμα Οπότε θα πρέπει πρώτα απ' όλα ρόλο να παίξει η ευρωστία της νομοθεσίας. Εάν γι' αυτό το λόγο καθυστερήσουμε λίγο, καλύτερα να καθυστερήσουμε λίγο και να έχουμε πιο σωστή νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η συγγήτρια για την ομάδα των φιλελευθέρων. Έτσι λοιπόν θα μιλήσω τώρα ως Κιώδης ε, η συγγήτρια. Και θέλω να ευχαριστήσω τον ε, Οτμάρ για όλο το, το έργο και επειδή ξεκίνησε ε, πολύ νωρίς να δίναμε κάποιους πιθανούς ενδυνάμεις συμβασμούς που καλώς ορίζουμε σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Κατανοώ την ανάγκη να προσπαθήσουμε και να μείνουμε στο φιλόδοξο και ταχύχρονο διάγραμμα. Και τώρα ως πρόεδρος μπορώ να πω ότι στη γραμματεία ε, εμείς ε, προσπαθούμε ε, να οργανώσουμε το χρονοδιάγραμμα και να δούμε και πιθανές ημερομηνίε για την υλοποίηση του τριμερούς διαλόγου που να ταιριάζουν με το χρονοδιάγραμμα αυτό. Τώρα, και πάλι υπό το ρόλο της κιόδους εισηγήτριας, για τους φιλελευθέρους να πω ότι δεν πρέπει να πάμε τόσο γρήγορα, ώστε να μην ε, υιοθετήσουμε κάποιες νέες ιδέες ε, που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοι και φυσικά ε, έχω και κάποιες ιδέες δικές μου που θα τις αναφέρω τώρα. Καταρχήν, παρουσίασα την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γενική απέτηση για σχέδια ε, επίλυσης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύνδεσμο με τέτοια σχέδια στις κεφαλαϊκές απαιτήσει, στη σχετική οδηγία των κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις οντότητες και ο ρόλος της EBA, της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Τραπεζών, που δόθηκε στον κανονισμό για την MBA θα πρέπει να είναι ότι συμμετέχει στο συντονισμό. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αν έχουμε ένα εθνικό σχέδιο πύληση, πρέπει να έχει ένα ρόλο διαφορετικά πώ θα γίνει ο συντονισμό. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζω το ότι δεχτήκατε ε, την ιδέα του διασυνοριακού, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε κάτι πιο γενικό. Δεν θέτω απαιτήσει ε, για ταμεία ή για κάποιε λεπτομέρειε, για εργαλεία, γιατί θα δώσει αυτό ε, στο Συμβούλιο την ε, δυνατότητα ε, να καθυστερήσει. Όμως, ε, αν υπάρχει ένα καλό σχέδιο, τότε μπορεί να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να υπάρχει απαλλαγή. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την πρόταση των πρασίνων, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να είναι αντί ε, του να έχουμε κάποιε απαιτήσει. Όσο ό,τι αφορά τους ε, μακροπροβλητικού ελέγχου, το έχω βάλει αυτό στο άρθρο 112 για την οδηγία. Ξέρω ότι ε, εσείς το εξετάζετε στο άρθρο του 443 στον κανονισμό. Ελπίζω να δείτε τι πρότεινα και εγώ, γιατί όπου και αν είναι, ορισμένοι από τους μηχανισμούς ε, που προτείνω, ξεκολουθώ να πιστεύω ότι θα είναι σκόπιμοι και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια απαγόρευση από την Κομισιόν, θέλετε. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι πρέπει να είναι μετά το γεγονό και όχι πριν. Στην πράξη δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη ευελιξία ε, για να μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί αυτό και ε, αν ε, η Κομισιόν θεωρήσει ότι πρέπει να το σταματήσει, τότε πρέπει να το κάνει στην πράξη και ίσως θα πρέπει να δώσει μια ειδοποίηση, μια προειδοποίηση μόλις ειδοποιηθεί. Δεν ε, ξέρω πώς η Κομισιόν θα κάνει αυτή την εποπτεία είναι ενδιαφέρον ε, το ότι προτείνεται να είναι μια κοινή απόφαση χρησιμοποιώντας και το κολέγιο, το συλλογικό σώμα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να θετήσουμε κι αλλού εκεί όπου υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Όμως ε, νομίζω ότι με μια κοινή απόφαση τελικά η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι αυτή που αποφασίζει. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτό συνάδει με τη γενική ε, κατεύθυνση που ακολουθεί αυτή η Επιτροπή. Κάποια άλλα τώρα θέματα που θέλω να σχολιάσω. Έχω παρουσιάσει κάποιες προτάσεις ε, για το benchmarking και για τα χαρτοφυλάκια που θα μπορούσαν ε, να είναι αντικείμενα διαχείριση μέσω διαφορετικών ε, τραπεζικών μοντέλων. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντική εξέλιξη, γιατί σε διεθνέ επίπεδο αναπτύσσονται αυτά τα χαρτοφυλάκια, αλλά ήδη η Ευρωπαϊκή Έρχη Τραπεζών το πράττει και στι ΗΠΑ και στην Ασία, και αυτό είναι από του τρόπου με του οποίου μπορούμε να έχουμε συγκρισιμότητα από περιφέρεια σε περιφέρεια. Έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα ε, σε σχέση με τις διαφορές, ε, με ε, την αναλογία μόχλευσης ή την αναλογία κεφαλαίου και benchmarking θα ξεκολουθούμε να έχουμε προβλήματα. Έτσι λοιπόν, λοιπόν είμαι υπέρ αυτού. Και επίσης και σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών. Θέλω να δείτε την τροπολογία με 770 για το θέμα αυτό, ώρες ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι ο συμβασμός που προτείνεται οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Εγώ έβαλα την ε, πρόταση ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια δυνατότητα ε, να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι οντότητες ε, στη μαύρη λίστα όταν υπάρχουν μια αρμοζή συμπεριφορές. Δεν θέλουμε να υπάρχει μετακίνηση από χώρα σε χώρα. Και επίσης ε, προτείνω ότι οι εξαγορές ε, των ε, συμβάσεων να υπόκεινται στις ίδιες διευθετήσεις clawback όπως και άλλα είδη πληρωμών bonus και ξέρω ότι το έχετε συμπεριλάβει αυτό στην πρότασή σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και θα ήθελα τώρα να περάσω στο πακέτο ανάπτυξης. Δύο σκέλη έχουμε εδώ. Το ένα το αναφέρατε. Καταρχήν για τις μικρές ε, και μεσές επιχειρήσεις. Εγώ θα ήθελα να δω ε, αλλαγή στη στάθμιση κινδύνου, αλλά προτείνω και έναν άλλο μηχανισμό που είναι ε, πρόσθετος, όχι αντί κάποιου άλλου. Δηλαδή να λέμε ότι θα έπρεπε να έχουμε απομόνωση ενός ποσού κεφαλαίου για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Αυτό δεν αρέσει τι τράπεζε, αλλά θεωρούμε ότι θα έχει νόημα γιατί θα τις αναγκάσουμε να έχουν ε, κάποιο συγκεκριμένο κεφαλαίο ή να ε, κάνουν προ το δανεισμό. Δεν ε, θέτω εγώ θέμα εποπτεία εδώ. Θα μπορούσαμε να έχουμε και μια προσέγγιση EBA, θα ήταν επιθυμητό, αλλά σα παρακαλώ να το εξετάσετε αυτό, γιατί είχαμε κάποιες εμπειρίες με τη στάθμιση κινδύνου και τη μείωσή τη και δεν αύξησε σε το δανεισμό. Στην Ιταλία λόγω έτσι λοιπόν ε, θα μπορούσαμε να βρούμε έναν άλλο μηχανισμό που να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει. Το άλλο τμήμα του πακέτου ανάπτυξης και εσείς έχετε θέσει κάποιες τροπολογίες για την χρηματοδότηση του εμπορίου και εγώ συμπλήρωσα αυτό το πακέτο θέτοντας κάποιες τροπολογίες που προσαρμόζουν ε, τα ανοίγματα και κάποιες τροπολογίες σε σχέση με τη ρευστότητα που έχουν να κάνουν με αυτό το πακέτο χρηματοδότησης ε, εμπορίου και νομίζω ότι συνολικά θα ήταν ε, πολύ καλές για την ε, προώθηση της ανάπτυξης παντού και κάτι τέτοιο θα ωφελούσε και εμάς φυσικά στην Ευρώπη. Αλλά οι τραπεζές μας είναι υπεύθυνε για μεγάλο βαθμό χρηματοδότησης εμπορίου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σχετικό αυτό το θέμα και νομίζω ότι σε διεθνές επίπεδο τώρα αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Κάποια άλλα σημεία που θα ήθελα να αναφέρω ε, σε διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους. Έχω συμπεριλάβει την ιδέα ότι δεν μπορεί κάποιος ε, να εξαιρέσει τον εαυτό του από τις απαιτήσει ε, δημοσιοποίησης με έναν τρόπο που δεν θα σεβόμαστε την δημοσιονομική σταθερότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό να το συμπεριλάβουμε Επίσης, ε, πρέπει να αξιολογηθούν ε, τα ρευστά διαθέσιμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανησύχησα ότι ένας από τους όρους της ρευστότητας ε, ήταν απλό ότι θα μπορούσε να κάνει κάποιος μια επαναγορά, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ τραπεζών, να ανταλλάξουμε τα περισσότερα μας στοιχεία. Δεν είναι ο είδος τουρισμού που θα ήθελα εγώ. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε κάτι πιο αυστηρό, ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια απλή ποικιλία διαθεσιμών σε μια εγκεκριμένη αγορά. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπό, αλλά καθώ ε, τώρα έχουμε πιο εξωτικέ ε, τέτοιε αγορέ αυπληρώμων καλό θα ήταν να το ορίσουμε αυτό. Και θέλω να πιστήσω την προσοχή σα και στην τροπολογία μου 600 για τη στρατηγική καταπολέμηση τη απάτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδιώκουμε μια τέτοια στρατηγική καταπολέμηση τη απάτη. Υποστηρίζω την ιδέα να μετακινηθούμε λίγο παρατερά για τη στάθμιση κινδύνου του δημοσίου χρέους παρά να ζητάμε εκθέσεις. Συμφωνώ ότι πρέπει ε, να αποτύχουμε κάτι προκυκλικό αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δείχνουμε ποιες είναι οι κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουμε κάτι άλλο πέρα από το μηδέν. Δεν μου αρέσουν οι εξισώσεις ε, με μηδέν στο κάτω μέρος, δηλαδή σημαίνει κάποιο ότι, πρέπει ότι μπορεί να επενδύει επάπειρον. Έτσι λοιπόν, ε, αν στη στάθμιση κινδύνου ε, κάτι σε σχέση με την ορίμανση. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια ισορροπία. Υπάρχει η ισορροπία στο Κοινοβούλιο που μπορούμε να κάνουμε με την ε, αναλογία, τη σταθερή αναλογία χρηματοδότησης. Ε, αυτό είναι πολύ σχετικό το θέμα. Ε, τώρα, για το ε, ε, θέμα της Βασιλείας 1 και το σχετικό κατώτερο επίπεδο, δεν νομίζω ότι πρέπει να το διαγράψουμε αυτό. Αν, ε, παραδείγματο χάρη, κάποιος έχει ένα χαρτοφυλάκιο για ένα ετός, μπορεί να άρει ίσως ε, το κατώτερο όριο της Βασιλείας 1, αλλά εγώ δεν θα ήθελα κάποιο άλλο μέσο να το αντικαταστήσει αυτό και επίσης θέλω συνέπεια με όσα κάναμε στην ε, EMEA και μπορώ να υποστηρίξω μια σταδιακή προσέγγιση σε στρώματα όπως προτάθηκε από τους Πρασίνους αλλά δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε ένα στρώμα τραπεζών που δεν πρέπει να επακούν τους κανόνες. Δηλαδή υποτίθεται ότι αυτοί οι κανόνες ε, είναι πολύ ισχυροί για όλες τις τράπεζες και ιδιαίτερα ισχυροί και αυστηροί για τις μεγάλες τράπεζες. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Και επόμενος ομιλητής, η Βίκη. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Πραγματικά καλωσορίζω τη διάθεση του εισηγητή να καταλήξουμε σε αυτό το πακέτο μέτρων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή όσο το δυνατόν γοργότερα και να προχωρήσουμε και μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα θα ε, δώσω τη διασφάλιση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι μεγάλη η πρόκληση. Γνωρίζουμε επίσης ότι πολλές, ε, πολλά προβλήματα ε, συναρτώνται με τις λεπτομέρειες και συμφωνώ και με τον εισηγητή ότι πρέπει μέσα στην ενιαία εσωτερική αγορά που πρέπει να διασφαλίσουμε με ισοδίκαιο πλαίσιο να λειτουργήσουν αυτά. Τίποτα δεν υπονομεύει περισσότερα την ενιαία εσωτερική αγορά από ότι κάποιες παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις και κάποιοι θα, ε, που ε, ε, εποφελούνται από κάποιες ξεχωριστές διατάξεις υπονομεύουν την ενιαία εσωτερική αγορά. Είναι κρίσιμη συγκέρια σημασία να διασφαλίζεται ένα τέτοιο γενικό πλαίσιο για όλους και να υπάρξει η ανάπτυξη μέτρων εμπιστοσύνης μέσα από αυτά και η οικονομική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει. Και πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε εκείνες ε, τις ε, ε, απαιτήσει χωρίς να τις αποδυναμώσουμε για να προχωρήσουμε και να υπάρχει και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ένα κοινό πλαίσιο. Πρέπει όμως να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν διαφορές στις εθνικές αγορές και στο παρελθόν αντιμετωπίζουν θέματα παρόμοια όπως αυτό αυτής της αναγνωρίζαμε ότι υπάρχουν διαφορές στις εσωτερικές ε, ε, διατάξεις που έχουμε στις αγορές μας, δίνοντας ένα πλαίσιο και περιθώριο στα κράτη-μέλη αναφερόμενοι στις ε, ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες ε, και τους όρους ε, και προϋποθέσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο εθνικό πλαίσιο. Αυτό είναι δυσκολότερο σε σχέση με έναν κανονισμό. Για, για παράδειγμα, σε σχέση με την συμφωνία όσον αφορά τη Βασιλεία 1 για τα ενυπόθηκα δάνεια και τις εγγυήσεις και σε σχέση με τις ε, διασφαλίσεις, ε, σε σχέση με κάθε χώρα και κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του ενίου πλαισίου, να δούμε σε λεπτομέρειες ε, τι ξεκινάμε και να μην καταλήξουμε με ένα πακέτο βασιλείας που θα λέει στον τίτλο ή στο, ας το στην επιφάνεια θα αναφέρει ένα ενίο πλαίσιο, όμως στις λεπτομέρειες δεν θα λαμβάνονται αυτά υπόψη. Το άλλο σημείο είναι να δούμε την παγκόσμια μεταρρύθμιση σε σχέση με τις 27 χώρες μέλη. Δεν θα πρέπει εδώ να ε, ακολουθήσουμε τον ρυθμό των βραδύτερων ή τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αν κάποιες χώρες θέλουν να πορευθούν ταχύτερα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ευελιξίας για να μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Χρειάζεται ταχύτητα και ρυθμός. Θα πρέπει να είμαστε όμως ιδιαίτερα ε, προσεκτικοί όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις μιας τέτοιας προσέγγισης. Αν αποφασίσει ένα κράτος μέλος να ακολουθεί ακολουθήσει μια ξεχωριστή ταχύτερη πορεία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις και σε άλλα κράτη. Συμφωνώ με πολλά που, ανέφερε ο εισηγητή ε, για την ανάγκη να δούμε τις εθνικές διαφορές. Όμως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δούμε σε σχέση με την εποπτεία τι θα μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να δούμε πιο ε, δημιουργικά τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τα κράτη-μέλη και για την αναγνώριση και εντοπισμό του συστημικού κινδύνου. Πρέπει να ενδυναμώσουμε την δυνατότητα να λαμβάνονται οι αναγκαίες αποφάσεις όσον αφορά διασυνοριακές τέτοιες συναλλαγές. Είναι πρόκληση το να αντιμετωπιστεί η ε, κατάσταση αυτή και πρέπει έγκαιρα να αντιμετωπίζεται προτού υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε μια άλλη χώρα και πρέπει φυσικά να λαμβάνονται υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες. Θα έλεγα ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν αυτά να λειτουργήσουν σωστά και στον κανονισμό και στην οδηγία για τα μακροοικονομικά εργαλεία, η μέσα και τις, ε, ε, τη λειτουργία τους. Κύρια σημασία για μένα έχει η κυριότητα τη σημασία η διαφάνεια. Και αυτό αφορά πολλές από τις τροπολογίες με τους στόχους που έχουν. Για τα κεφάλαια θα έπρεπε να μπορέσουμε να ε, δούμε τις ανάγκες όσον αφορά και τις, τα τις μετοχές, τα μερίδια, πρέπει να εξεταστούν και οι συνεταιρισμοί με τις ιδιομορφίες τους και σε σχέση με τροπολογίες και από το ΕΛΚ και τους σοσιαλδημοκράτες με, που είναι συναφείς μεταξύ τους, θα πρέπει να δούμε και την αναλογία κεφαλαίων. Πρέπει να υπάρχει πραγματική διαφάνεια που θα διασφαλίζεται και σωστή εποπτεία για την ε, λειτουργικότητα όλων αυτών. Αυτό αφορά και τα μειοψηφικά ε, δικαιώματα μειοψηφίας μεριδιούχων για την ε, φερεγγιότητα, τη ρευστότητα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το LCR θα μπορεί ως πράξη κατ' εντολήν κατ' εντολήν ε, δράση να αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν όμως ε, και ε, θέματα που αφορούν τους βιομηχανικούς και επιχειρησιακούς κύκλους. Ξέρω ότι η Επιτροπή Βασιλείας εξετάζει και εργάζεται επί αυτών των λεπτομεριακών θεμάτων. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ευθυγραμμιστούν αυτά τα συμπεράσματα σε σχέση με τις συστάσεις της Επιτροπής Βασιλείας το συζήτησαν οι τράπεζες και νομίζω ότι μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν πραγματικά ε, σωστή για την, ε, ε, τις αναλογίες μέχρι, τον Ιανουάριο που θα μπορούσε να γίνει αυτό. Είναι κέρια σημασία να το πετύχουμε για να αποφύγουμε επανάληψη φαινομένων τέτοιων κρίσεων όπως αυτές που ζήσαμε στο παρελθόν και για τη διασφάλιση της ε, ρευστότητας κυρίως όσον αφορά και χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης, κέντρο-ανατολικό ευρωπαϊκών χωρών, θέματα ρευστότητας που πρέπει να αντιμετωπιστούν και σε σχέση με τις τράπεζές τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένα συντονισμός πρέπει να διασφαλίζεται για να είμαστε πιο λειτουργικοί. Από την άλλη πλευρά κάποιες τροπολογίες θέλουν να αποδυναμώσουν ή να παμβλύνουν τα κριτήρια για την ε, ρευστότητα και υπάρχουν και ίσως υπερβολές. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλα αυτά τα θέματα, να υπάρχει η ελαστικότητα σε σχέση με την περίοδο, τη μεταβατική περίοδο εποπτείας, αλλά πρέπει όμως το μήνυμα που θα αποστείλουμε να είναι στεναρό και ισχυρό ότι δεσμευόμαστε όσον αφορά αυστηρές προδιαγραφές για τη ρευστότητα, για τη μόχλευση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι Πέντε χρόνια πέρασαν από τότε που ξέσπασε η κρίση σε σχέση με τις ε, υπηρεσίες στον χρηματοοικονομικό τομέα και η μόχλευση ήταν ένα σημείο κλειδί ε, που είχε σημασία ιδιαίτερη. Θα πρέπει να δούμε το, <clears throat> την ανάγκη να υπάρξει διαφάνεια και θα πρέπει να μπορέσουμε να επεξηγήσουμε πώς διαφορετικά πρότυπα μπορούν να επιτύχουν διαφορετικό επίπεδο μόχλευσης. Χρειάζεται δέσμευση για την εισαγωγή αυτού του ε, στόχου κατανοώ την διαφοροποίηση διαφορετικών προτύπων προσέγγισης και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε διατυπώσεις που θα ε, τύχουν κοινή συνένεση ε, και από πλευρά ε, των μελών που ζητούν ως ευρωβουλευτές να είναι δεσμευτικά αυτά τα πρότυπα μόχλευσης ιδιαίτερο μέλημα θα πρέπει να είναι να μειωθεί το επίπεδο κινδύνων στο οποίο εκτίθενται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μπορέσουμε να, είμαστε, ε, υποστη, να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνώ με αυτό. Πολύ καλή δουλειά σε πολλούς τομείς ε, έγινε σε σχέση και με την τροπολογία μου 856 όπου ε, σε σχέση με ε, θέματα για τυποποιημένες ε, διαδικασίες ε, που θα πρέπει να εισαχθούν, εξετάζονται. Θα ήθελα να υπάρχει και μικρότερος κίνδυνος όσον αφορά και την χρηματοδότηση έργων που θα στοχεύουν στις υποδομές. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην χρηματοδότηση προγραμμάτων και σχεδίων που λειτουργούν και υπό την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα πρέπει να δούμε και το σχέδιο των Project Bonds Initiative την πρωτοβουλία ομολόγων έργου, ευρωομολόγων εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο χρηματοδότησης πρέπει να δούμε και τις λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν υποστηρίζω όμως το θέμα της ε, ε δανειοδότησης ε, εμπορευματικής δράσης, εμπορικής δράσης όσον αφορά ενυπόθηκα δάνεια και στεγαστικές πολιτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με το επίπεδο μόχλευσης ε, και τα αρνητικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στο ε, παρελθόν. Θα πρέπει να προστατευτούμε έναντι προβλημάτων που ελοχεύουν όσον αφορά ε, μια τέτοια προσέγγιση. Ιδιαίτερα όσον αφορά το πλαίσιο Βασιλείας 2. Ε, Ιδίω υποστηρίζω την πρωτοβουλία των αυστηρών βέλτιστων προδιαγραφών δράσης, benchmark ε, initiatives. Και για την διαφάνεια όπου είπα ότι έχει ιδιαίτερη σημασία υπάρχουν πολλές τροπολογίες και ιδιαίτερα όσον αφορά τις αλλαγές που θα πρέπει να διασφαλίσουμε ασφαλή μέθοδο δραστη, δράσης και δραστηριοποίησης ε, ε, έναντι για παράδειγμα των ε, επενδυτών ή εκείνων που επενδύουν τις καταθέσεις τους σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Όσον αφορά τις, τον τομέα ασφαλιών μεριδι, αγοράς μεριδίων μετοχών ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι καταθέτες δεν θα ε, δουν ότι απασφαλίζονται τα κονδύλια τους ε, για χρήση, αδιάκριτη χρήση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ευχαριστώ για τις ε, συμβιβαστικές ε, τροπολογίες και την ε, διάθεσή σας να δεχθείτε προτάσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τις διακοιμάσεις, όσον αφορά το έμπερ και την σωστή επιλογή. Νομίζω ότι το εύρος δράσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά ε, το εταιρικό δίκαιο και να δούμε την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου είδα ότι πολλές ε, γυναίκες ήταν εκείνες ε, οι οποίες επομιζόντουσαν πολλές φορές πολλούς κινδύνους να ε, είναι κανείς πεισμένος ότι αν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες θα μειώνεται αυτόματα ο κίνδυνος δεν είναι δεδομένο. Και για τις αμοιβέ ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Αρλίν για το CRD3 Ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν υλοποιήσει τις προτάσεις και τις απαιτήσεις του CRD3 και θα πρέπει με την εκκίνηση αυτής της συζήτησης να διασφαλίσουμε ότι δεν θα απολεστεί το έργο που κάναμε κατά το παρελθόν και θα είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι αναφέρονται και διαφορετικές προσεγγίσεις σε τροπολογίες ευρωβουλευτών θα ήθελα όμως να μην υπάρχει διαρκώ ε, διαρκώς συσσόρευση ε, προτάσεων για εξαιρέσεις. Προσβλέπω στη στενή συνεργασία με τον ε, εισηγητή για την εξειδίκευση των προτάσεων σε σωστούς συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. Φιλίπ. Ευχαριστώ, Φιλίπ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Ότμαρ και τη Τζουλιά αλλά και όλα τα μέλη της ομάδας που εργάστηκαν σκληρά για να γράψουν αυτές τις τροπολογίες στην ε, διακεφαλαϊκών απαιτήσεων 4 και βεβαίω ε, δεν πρέπει να υποτιμούμε την ε, συνεισφορά του. Τώρα να ξεκινήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ότμαρ, συμφωνώ πως δεν πρέπει να καθυστερήσουμε χωρίς λόγο. Οπότε θα ήθελα να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αρκεί να έχουμε ποιοτική δουλειά και εγώ είμαι υπέρ του 80-20, δηλαδή καλύτερα να περάσουμε ένα 80% καλό παρά να περιμένουμε το, τελικό, ή το τελευταίο 20% που θα χρειαστεί άλλους 10 μήνες. Για μένα ο βασικός λόγος για να κινηθούμε γρήγορα είναι για να προλάβουμε το Συμβούλιο. Συμφωνώ με τον Σαμπόλε, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς εδώ πέρα πριν από το Συμβούλιο θα επηρεάσουμε. Εάν αργήσουμε θα είναι δύσκολο να αλλάξουμε τη θέση του Συμβουλίου. Οπότε υπ' αυτή την έννοια συμφωνώ να βιαστούμε. Από την άλλη, αν δούμε το πλαίσιο με τον, το 9% το οποίο απαιτείται ως κεφαλαιακή απέτηση την 1η Ιουλίου, φαίνεται πως δεν έχουμε χρόνο. Οπότε δεν θα έχουμε μεγάλη διαφορά εάν χρειαστούμε άλλους τέσσερις μήνες ε, παραπάνω. Δεν είναι τόσο πιεστική η κατάσταση ώστε να είμαστε τσαπατσούλιδες. Το βασικό λοιπόν είναι να προλάβουμε το Συμβούλιο. Όλα τα υπόλοιπα, για όλα τα υπόλοιπα είμαι ελαστικός. Δεν ε, καίγομαι τόσο πολύ ε, όσο παραδείγματο χάρη για την κρίση του ευρώ. Κατόπιν θα αναφέρω τέσσερα βασικά ζητήματα και θα συμφωνήσω με κάποιους συναδέλφους και θα ξεκινήσω από τις αμοιβέ και τα κίνητρα. Ειλικρινά έχω αρχίσει να βαριέμαι αυτό που μας λένε ε, ξέρετε αυτό είναι λαϊκισμός. Δεν συμφωνώ. Γιατί εάν ζητάμε από τον κόσμο στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στη Γαλλία οικονομία με την έννοια ότι η μισθή πρέπει να είναι ανάλογη με την παραγωγικότητα, κανείς ακόμα δεν μου έχει δώσει επιστημονικά στοιχεία το, για το ότι τα επίπεδα των μισθών που βλέπουμε στην Deutsche Bank, στους General και λοιπούς ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε δημιουργία αξίας. Επίσης, εάν ε, υπήρχε επιστημονική σύνδεση ε, μεταξύ αυτών των μισθών ε, και, των, και της δημιουργίας αξίας, ε, τότε δηλαδή η Άγγελα Μέρκελ δεν δημιουργεί καμία αξία. Και εμείς εδώ πέρα, να το πω, θεωρώ πως δεν δημιουργούμε επίσης καμία αξία. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες που βασίζονται στην το οδηγία κεφαλαιακών αποτήσεων 3 και λέμε πως ε, ο μισθός, ε, ο κειμενόμενος, τα μπόνους δεν μπορεί να είναι πάνω από τον σταθερό. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δουλέψει με ποσοστά. Εγώ είχα δουλέψει μία χρονιά μόνο ε, τα κίνητρα ήταν παραπάνω από το βασικό μισθό. Αλλά για να είμαι δεν χρειάζομαι παραπάνω για κίνητρο. Μη μου λέει κανείς πως χρειάζεται πενταπλάσιο του μισθού του για να κινητοποιηθεί να κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι λάθος. Λάθος. Και εάν έχει κάποιο στοιχεία που το διαψεύδουν να τα δω. Αλλά δεν υπάρχουν. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Επίσης υπάρχει εδώ πέρα η ιδέα ενός maximum ε, το οποίο, maximum αμοιβή, το οποίο θα είναι ένας λόγος ε, επί 40, από το minimum έως το maximum. Και να αναφερθώ τώρα στα βασικά ζητήματα ρευστότητας, ε, μόχλευσης και επάρκειας. Και το βασικό θέμα εδώ πέρα είναι εάν όλοι θα έχουν τους ίδιους κανόνες, αλλά θα υπάρχει και επικοινία. Και εδώ πέρα συμφωνώ με τον Ότμαρ και με τους σκιώδεις ηγητές. Ξέρουμε πως ε, τα ίδια μέτρα για όλους δεν ε, λειτουργούν και γι' αυτό οι δεν θα εφαρμόσουν τη Βασιλεία 3 για όλους. Να εμείς θέλουμε, ναι εντάξει, αλλά τότε να κάνουμε διακρίσεις. Και λέμε πως κατά βάση υπάρχουν τρεις ε, κατηγορίες. Αφενός έχουμε τις εταιρείε τις παγκόσμια συστημικές που έχουμε ειδικού κανόνες. Κατόπιν, στο ασφαλές άκρο έχουμε ε, παραδοσιακές βασικές τράπεζες ε, όπως θέλετε πείτε τις που έχουν καταθέσεις και δίνουν δάνεια στην πραγματική οικονομία μπορεί να είναι μεγάλες και μικρές μπορεί να είναι συνεταιριστικές ε, μπορεί να είναι κανονικές αε εμείς λέμε πως είναι μια ξεχωριστή κατηγορία και πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε αυτές και μετά υπάρχει οτιδήποτε είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι πολλά. Λέμε λοιπόν πως θα κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε κεφάλαιο, μόχλευση, ρευστότητα, ε, τρία επίπεδα και τρεις κατηγορίες. Όπως και ο Ούντο είμαι διατεθειμένος να συζητήσω διαφορετικές κατατάξεις, ε, πρέπει να είμαστε απλοί. Όσο πιο περίπλοκη η νομοθεσία, τόσο πιο εύκολα παρακάμπτεται και νομίζω πως η σαφήνεια εδώ πέρα μας βοηθάει. Πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Είτε α, β, γ ή δ κατηγορία. Όχι να λέμε ναι, αλλά ε, είμαι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Όχι, ή το ένα είσαι ή το άλλο. Πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν αυτό. Και μόλις συμφωνήσουμε για τις διακρίσεις αυτές. Πρέπει να μιλήσουμε για τις ε, κεφαλαιακές ε, απαιτήσει. Ξέρετε πως είμαστε πιο φιλόδοξοι από τους Βρετανούς, ε, τις Βρετανικές ρυθμιστικές αρχές. Έχουμε πει ξεκάθαρα πως ε, θέλουμε μεταξύ 8 και 10 τις 100 για τις βασικές τράπεζες, 10 με 15 για την μεσαία κατηγορία και 16 με 20 για τις παγκόσμιες συστημικές, αλλά συμφωνώ και με τον Αγχέλ ε, Χουρία που ήρθε εδώ πέρα χτες. Ε, τι είπε, όχι να σταματήσουμε αυτές τις λακίες, χρειαζόμαστε υποχρεωτικά ποσοστά μόχλευσης, χρειάζονται, αλλιώς δεν γίνεται αλλιώς ε, η αξιολόγηση του κινδύνου, η στάθμιση του κινδύνου. Οπότε η ομορφιά εδώ πέρα είναι η απλότητα του συστήματος. Και πάλι λέμε για τη μόχλευση θα πρέπει να έχουμε 2 με 3% για τις ε, βασικές τράπεζες, 9 ε, με 10% για τις παγκόσμιες και 6% ε, για το ενδιάμεσο. Και αυτά δεσμευτικά. Για τα υπόλοιπα συμφωνώ με την Σάρων για το πώς θα κάνουμε πιο περιοριστικούς τους ορισμούς δεν μου αρέσουν αυτή τη στιγμή και θα θέλαμε να κάνουμε κάτι και με το SFR. Θεωρώ πως εδώ πέρα δεν είμαστε η μόνη ομάδα που το θεωρεί αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό. Κάτι άλλο που ξέρουμε πως απασχολεί την ε, Κομισιόν και θα μπορούσαμε να δούμε εδώ πέρα ως έναν βαθμό αυτό το shadow banking. Δεν είναι το θέμα ότι η Κομισιόν σκέφτεται να κάνει κάτι και άρα εμείς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κανονισμό για να κάνουμε κάτι. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε αυτό το κείμενο είναι να διαχειριστούμε τις ροές χρημάτων, να δούμε τις ροές χρημάτων μεταξύ τραπεζών που ρυθμίζουμε και λοιπόν. Και εκεί πέρα το να παίξουμε με το ποσοστό ρευστότητας και με πιθανά πλαφών στις ε, ροές ε, τις χρηματικές μεταξύ τραπεζών ρυθμιζόμενων και μη θα μας επιτρέψει τουλάχιστον σταδιακά να κόψουμε τη χρηματοδότηση στις σκιώδεις αυτές τράπεζες. Με, ε, έτσι θα τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Και σε τελική αναλύση δεν θέλουμε σκιώδεις τράπεζες. Αυτή, ε, αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Ε, αντιλαμβάνομαι πως ο εισηγητής ε, έχει κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ είμαι και έτοιμος να ψηφίσω και αύριο. αν δεχτεί τις τροπολογίες μας ο εισηγητής βεβαίως. εντάξει δεν θα γίνει. Ωραία εντάξει. Εμείς είμαστε διεθνείς λοιπόν να συνεργαστούμε, να κινηθούμε γρήγορα, αλλά αυτό εξαρτάται από τη, τη φύση των συμβιβαστικών προτάσεων που θα δούμε. Θα σταματήσω εδώ. Δεν χρησιμοποίησα τα 12 λεπτά που εξάντλησαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Γιούργεν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, για το χρονοδιάγραμμα. Με αυτό να ξεκινήσω. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία και υποστήριξη. Το τονίζω αυτό. Υπήρχε πάρα πολλή δουλειά που έπρεπε να γίνει και ήταν πολύ καλή αυτή η συνεργασία. Για το χρονοδιάγραμμα το υποστηρίζουμε να πάμε γρήγορα αν γίνεται. Καμιά φορά έχω και επιφυλάξει όταν βλέπω πόσα πράγματα εντάσσονται στο πρόγραμμα και υποχρεώσει. Πρέπει να δούμε πώ θα τα καταφέρουμε λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα. Καταρχήν επί των τροπολογιών κυριότερους πυρήνες έχουμε που προσπαθήσαμε να, εντάξουν, να ενταχθούν και τα όσα αναφέρθηκαν νομίζω δείχνουν ότι είναι συμβατά, πρέπει να υπάρχει συμβατότητα. Το πρώτο, διατήρηση μιας ε, αποκεντρωμένης διαχείρισης όσον αφορά τις τράπεζες. Ε, το Κλασικό τομέα τομέας δραστηριοποίηση των τραπεζών που θέλουμε να ενδυναμωθεί και για τις μελλοντικές κρίσεις να αποφύγουμε φαινόμενα όπως στο παρελθόν. Να αποφύγουμε κυρίως οι φορολογούμενοι να κληθούν να πληρώσουν τα σπασμένα. Για το θέμα των ιδίων κεφαλαίων ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια η ομάδα πραγματογνωμόνων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας τοποθετήθηκε για το 20% το οποίο θα μπορούσε να είναι εφικτό και σύμφωνα με αυτή την πρόταση και εμείς όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, υστερότερα έγινε αυτό, αλλά και εμείς τοποθετηθήκαμε υπέρ μιας μεγαλύτερης κεφαλαιακής υποχρέωση ε, υποχρέωσης και έχουμε και τροπολογία προς αυτό το στόχο. Αν υπάρξουν προβλήματα με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα επανακεφαλαιοποίησης, ανακεφαλαιοποίησης ε, τραπεζών. Πιστεύουμε ότι η ΕΒΑ μέσω ενός προγράμματος για περιπτώσεις κρίσεων πρέπει να καθορίζει ποια, ποια είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Είναι θέμα και ορισμών ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σωστές διαφοροποιήσεις, σωστά όρια. Για το θέμα της ε, ρευστότητας και το funding ratio για την αναλογική κεφαλαίων Πιστεύουμε ότι πρέπει από το 2018 να είναι δεσμευτικό αυτό και για τη ΣΕΣΙΑ πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση κατά 100% ως ποσοστό θα πρέπει να ε, μην επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας. Για το leverage ratio, το ποσοστό μόχλευσης, έχουμε συζητήσει επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα τα ταμιευτήρια, δεν είναι χωρίς προβλήματα μια τέτοια πρόταση. Όμως πιστεύουμε γενικότερα ότι αυτή η πρόταση πρέπει να υποστηριχθεί από πλευράς μας και το δυνατόν πιο σύντομα πρέπει να υλοποιηθεί ώστε να μπορεί να λειτουργήσει το 2016. Νομίζουμε ότι είναι το πιο σκόπιμο μέσο, <clears throat> το πιο αποτελεσματικό μέσο σε σχέση με την αντιμετώπιση κινδύνων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι μια κλιμακούμενη προσέγγιση πρέπει να λειτουργήσει που θα λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά πρότυπα επιχειρησιακά πρότυπα. Είμαστε σε συζήτηση με ταμιευτήρια, με συνεταιριστικές τράπεζες και θα πρέπει να μπορέσει με τέτοιο τρόπο να διαφοροποιηθεί η προσέγγιση ώστε οι ανάγκες τους να καλυφθούν όσον αφορά και την ε, συμμετοχή τους ε, σε δημόσιες προμήθειες ε, και συμβάσεις και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το επίπεδο τράπεζες, τα ιδρύματα δηλαδή χρηματοπιστωτικά που θα εντασσόντουσαν σε αυτό το πλαίσιο. Και κατά τα άλλα θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα σε αυτό το οποίο ο εισηγητής πρότεινε για κάποιες τοπολογίες. Απορρέει από τα όσα προανέφερα η προσέγγιση του single rule ε, που περιορισμένα υποστηρίζεται διότι πιστεύουμε ότι μικρότερες τράπεζες, ε, ταμιευτήρια, συνεταιριστικοί τέτοιοι ταμιευτικοί οργανισμοί θα μπορούσαν να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις. Το τονίζω αυτό πρέπει πιο διαφοροποιημένα να ληφθούν οι ανάγκες τους υπόψη χαιρετίζουμε την προσέγγιση να έχουν την δυνατότητα οι εθνικές αρχές να προσαρμόζονται όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες τους. Θα το υποστηρίζαμε αυτό. Για τις άλλες τροπολογίες, πολύ σύντομα, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει σε πολλά θέματα ευρύτερη συνένεση και υπάρχουν και πολλές τροπολογίες που πιστεύουμε ότι είναι σωστές και που ενδιαφέρουν ενδιαφέρουσες προτάσεις υποβάλλουν και θα μπορούσαμε να τις υποστηρίξουμε. Στους πρασίνους ενδιαφέρον βρίσκουμε την προσέγγιση, ενδιαφέρουσα την προσέγγιση την η ιδιαίτερη πρόθεση κλασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων και να δούμε το πώς ε, από πλευράς ε, των αριστερών κάτι τέτοιο ήταν ένα αίτημα στην ε, Ομοσπονδιακή Γερμανία και η εισαγωγή ενός δεσμευτικού ποσοστού μόχλευσης και με ένα κλιμακούμενο πρότυπο που θα μπορούσε ίσως να έχει θετικές επιπτώσεις. Η ιδέα των ALDE, της ALDE για το benchmarking, τις βέλτιστες προδιαγραφές προτύπων κινδύνου και αυτό φαίνεται ότι είναι κάτι το λογικό για την στάθμιση των ε, κινδύνων είχαμε κριτική φωνή τοποθετηθεί ε, από αυτού. Από την μία πλευρά είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει καμία δραστηρι... κανένα επίπεδο χωρίς κινδύνους στην καθημερινή ζωή. Απ' την άλλη πλευρά όμως όταν σταθμίζουμε υψηλότερα κάποιους κινδύνους όσον αφορά τις ε, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση. Επιβάρυνση που τουλάχιστον σε σχέση με κάποια κράτη-μέλη δημιουργούν πιέσεις ε, όσον αφορά και τις, ε, τον τομέα των δαπανών. Αν κάτι τέτοιο είναι σκόπιμο, νομίζουμε ότι ε, μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Θα πρέπει πολύ προσεκτικά και συνετά να δράσουμε για όλα αυτά. Αυτά εν συντομία. Πολλά αναφέρθηκαν από τους άλλους συναδέλφους. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω αυτά. Και γι' αυτό επαρκούμε σε αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Έχω πολλούς ομιλητές από το ΕΛΚ. Θα ακούσουμε δύο-τρεις και κατόπιν έναν από τους σοσιαλιστές, έναν από τους ελεύθερους και να κάνουμε μια τέτοια περιτροπή. Ζαν πολύ καταρχήν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, Πρόεδρε, για να μπορούν όλοι να μιλήσουν ε, στο χρόνο που είναι επόμενοι. Καλύτερα να μιλήσουμε 12 λεπτά. Θα μιλήσω για γενικά θέματα γιατί πίσω από αυτή τη ρύθμιση θα πρέπει να δούμε τα οικονομικά συζητήματα. Καταρχήν, ε, η συζήτηση που γίνεται τώρα δημιουργεί κάποιες ε, ταραχές ε, στο βαθμό που οι αγορές ε, ήδη βλέπουν τις τράπεζες ε, σαν να έπρεπε να σέβονται τους κανόνες που δεν έχουν καθοριστεί ακόμη. Έχουμε ουσιαστικά ε, τη σιγουριά ότι η Βασιλεία 3 δεν θα εφαρμοστεί στις ΗΠΑ και ταυτόχρονα απαιτούμε από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες σε πολύ αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα ή τη φαραγκαιότητα. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή ε, πολύ ειλικρινά πέρα από τη συνηθισμένη διατύπωση κάνει πολύ καλή δουλειά και πραγματικά με κέρδισε και στις τροπολογίες. Από ό,τι είχα εγώ σε άλλη έτσι λοιπόν συγχαρητήρια και κουράγιο για να συνεχίσετε αυτή την αξιόλογη δουλειά. Για κάποια σημεία μόνο τώρα θέλω να αναφερθώ. Για το πρόβλημα των σύφης ε, ε, νομίζω ότι δεν ε, πρέπει να επιταχύνουμε τις απαιτήσει. Έχει προβλεφθεί για το 2016 γιατί διαφορετικά αν το απαιτήσουμε για το 2013 θα βάλουμε αυτά τα ιδρύματα σε πολύ δύσκολη κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Τώρα σε ό,τι αφορά τον λόγο της φεργιότητας, νομίζω εδώ πρέπει να δούμε τι έχουμε στην οδηγία ε, για τους ε, ομίλους, χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Επίσης ε, πρέπει να μην έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού σε σχέση με τη μόχλευση στην Ευρώπη. Είναι προβληματικό το θέμα της μόχλευσης και ε, σήμερα δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα, κυρίως για τους λόγους που ανέφερα, σε σχέση με την εκτίμηση που κάνουν οι αγορές για την εικονότητα των τραπεζών σε, πολλά χρόνια, σε κάποια χρόνια να σεβαστούν κάποιες απαιτήσει που δεν είναι γνωστές ακόμα. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, το άρθρο 404, ε, εκεί ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ο εισηγητής πρέπει να σκοπεύει σε λήψη ρεαλιστικών μέτρων για τα θέματα τώρα που πρέπει ε, να τα δούμε περισσότερο. Πρέπει να δούμε το θέμα της πελετίας και το ορισμό της πελατείας. Επίσης, ε, ήθελα κλείνοντας να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη τις πτυχές ε, της συγκεκριμένης λειτουργίας των τραπεζών. Ξέρω ότι κάποια κράτη θέλουν πιο αυστηρή νομοθεσία, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κατάλληλη εποπτεία. όμως πρέπει να είμαστε λογικοί εδώ, πρέπει να δώσουμε στους επόπτες ε, την κατάλληλη νομική βάση για να μπορούν να ασκούν ε, τις αρμοδιότητες ελέγχου και όχι να μπούμε σε μια υπερβολική ρύθμιση ε, και οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν όσα έγιναν στη Βασιλεία του στο G20 χωρίς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και σήμερα θέλουμε να ρυθμιστούν αυτά μέσω ευρωπαϊκής ρύθμισης. Όμως θα έπρεπε ίσως να τα σκεφτούμε λίγο νωρίτερα αυτά τα θέματα σε επίπεδο κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Ότμαρ στις αρχές του παρατηρήσεις. Εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδελφούς που το αποκαλούν διαφοροποίηση και όχι συγκεκριμενοποίηση. Θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη λοιπόν περισσότερο το γεγονός πως οι τράπεζες είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένες ε, στην Ευρώπη και εντός ε, κρατών μελών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη και Είμαστε βεβαίως ε, υπέρ ε, της εμβάθυνσης της ε, κοινή αγοράς. Στον τομέα των τραπεζικό και βεβαίως δεν θα πρέπει να οδηγήσουμε την Ευρώπη σε μια στασιμότητα. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα με χαμηλό κόστος για την οικονομία και αν το κάνουμε ε, όχι μόνο για τις ε, τράπεζες ε, της συστημικής σημασίας αλλά για ολόκληρο τον τομέα πρέπει να γίνουν κάποιες διακρίσεις και η διακρίση αυτή εάν βασίζεται σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό δεν μειώνει τις προσπάθειες εναρμόνισης οδηγίας και κανονισμού. Δεν είναι αντίθετη με ενιαίους κανόνες ή όπως αλλιώς το πείτε. Εγώ θα έλεγα μου πως με τη διαφοροποίηση αυτή μπορούμε να έχουμε ε, πραγματικά ίσους όρους ανταγωνισμού και το θέμα δεν είναι μόνο για τις ε, οικονομίες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης αλλά βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη πως σε αυτό το κομμάτι της Ευρώπης έχουμε ε, διαφορετικό χρηματοοικονομικό τομέα που τώρα δημιουργείται και έχει δεσμούς εξάρτησης με τράπεζες στην παλαιά λεγόμενη Ευρώπη και θα ξέρετε πως μόνο το τρίτο τρίμηνο πέρσι ε, έγινε ανάληψη 35 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις τράπεζες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε υπάρχουν προκλήσεις συγκεκριμένα για αυτές τις χώρες και για άλλες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις αλλά σαφώς ε, η δομή του τραπεζικού συστήματος εκεί με τις συνεταιριστικές τράπεζες που παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά όπως είπα πάλι αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ανατολική Ευρώπη. Και νομίζω λοιπόν πως ε, αυτή η διάκριση μπορεί να ενισχύσει αυτόν τον ε, κανονισμό και να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση του κανονισμού για να δημιουργήσουμε και ανάπτυξη και όχι να εμποδίσουμε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ Σάρων. Ευχαριστώ. Κάρεν. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κάρας για την εξαιρετική του προσέγγιση, η οποία είναι ανοιχτή απέναντι στους συναδέλφους. Ε, μάλιστα προσπαθεί να συνδυάσει την ποιότητα με την ταχύτητα. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα αυτό, το οποίο συζητάμε σήμερα και πρέπει να δώσουμε βεβαιότητα στις αγορές και στις τράπεζες ε, σε σχέση με την εφαρμογή της Βασιλείας ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε και την εμπιστοσύνη στον τραπεζικό μας τομέα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία θέματα. Καταρχήν, αυτό το Κοινοβουλίο έχει παράδοση τα τελευταία έτη να επιθυμεί να ενδυναμώσει τις αρμοδιότητες των Ευρωπαίων Εποπτών, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Συμφωνώ με τον Ότμαρ όταν λέει ότι η νομοθεσία είναι για τους νομοθέτες, δεν είναι για τους επόπτες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή συνεισφορά και στο επίπεδο 2 οι επόπτες θα πρέπει να θέτουν αρχές στην νομοθεσία, αλλά όταν μιλάμε για εποπτεία δεν μιλάμε αυτόματα για τις εθνικές εποπτικές αρχές. Εγώ έχω δει κάποιες ε, τροπολογίες που θέλουν να διευρύνουν ε, ε, τη δυνατότητα κριτικής ευκαιρίας για τους εθνικούς επόπτες και εγώ νομίζω ότι και εμείς ε, πριν να ξεκινήσουν ε, οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς να επιμείνουμε για αυτές τις αρμοδιότητες, της εξουσίες της EBA και της ESRB. Και ήδη υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία στην ε, έκθεσή σα. Είναι σημαντικό να έχουμε στους κανόνε για όλου, αλλά είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι και οι κίνδυνοι αξιολογούνται βάσει τη ίδια μεθόδου ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα ε, πρόβλεψης για την εφαρμογή της Βασιλείας 2 σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτό το θέμα επιμένω γιατί βλέπω να υπάρχουν αποκλίνουσες τροπολογίες. Έκανα κάποιες προτάσεις σε σχέση με την ενδυνάμωση της ε, θέσης του ESRB και τη θέση της CBA, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και επίσης ε, όταν υπάρχουν πρόσθετες ε, απαιτήσεις αντικυκλικού κεφαλαϊκού αποθέματος και ελπίζω να το διερευνήσετε αυτό, να το εξετάσετε προκειμένου να υπάρχει ενδυνάμωση, ενίσχυση. Το δεύτερο το θέμα της, ε, του λόγου ρευστότητας και το τι οθετούμε ως ρευστά διαθέσιμα. Εδώ θέλω να επιμείνω στην υψηλή ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, γιατί σε ορισμένε τροπολογίε μπορεί ε, κάποιο να δει ότι υπάρχει αποδυνάμωση του στοιχείου αυτού. Αλλά από την άλλη, όπως κάνει και η σημερινή νομοθετική πρόταση, παίρνουμε τη θέση ότι τα δημόσια ομόλογα θεωρούνται ως ρευστά διαθέσιμα και τα, οι τίτλοι, οι ευρωπαϊκοί τίτλοι που είναι σημαντικοί για την αγορά των υποθηκών δεν υιοθετούνται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ένα είναι υψηλή ποιότητα και το άλλο δεν είναι. Έτσι λοιπόν, εγώ στις ε, τροπολογίες μου υιοθέτησα ε, μια προσέγγιση σχετικά με αρχές που πρέπει να εκπονήσουμε, να εκπονήσουμε περαιτέρω στο επίπεδο 2 και από την EBA, όπου έχουμε πραγματικά κριτήρια ποιότητας ε, σε συνδυασμό με το κούρεμα και ελπίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε περαιτέρω στην προσέγγιση αυτή. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα πάντα φυσικά στον κανονισμό, αλλά μπορούμε να βάλουμε κάποιες αρχές ε, για να έχουμε μια ευρύτερη αξιολόγηση της, του τι είναι υψηλή ποιότητα. Και είμαι ανοιχτή να το συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα, αλλά είναι σημαντικό ζήτημα, τουλάχιστον για ορισμένα κράτη-μέλη, όπου έχουμε ε, μία ε, μεγάλη αγορά σε ό,τι αφορά τις υποθήκες σε συνδυασμό με πρόβλημα εξεύρυσης χρηματοδότησης. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω αφορά τη μόχλευση. Και συμφωνώ με την ε, πρότασή σας να περιμένουμε την περίοδο αξιολόγησης. Έχω θέσει κάποιες ε, τροπολογίες δυνάμει των οποίων κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη και η θέση των δημοσίων τραπεζών γιατί ε, ε, μπορεί να υπάρχει κίνδυνος ε, ε επιδείνωση θέσης θέση των τραπεζών αυτών. Δεν ζητώ εξαιρέσει, αλλά νομίζω ότι πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια τη αξιολόγηση και θεωρώ ότι είναι σημαντικό η θέση σε ισχύ ε, μάλλον η ημερομηνία θα ισχύσει να είναι η ίδια με την δημοσιοποίηση. Γιατί αν έχουμε διαφορετική ημερομηνία για την δημοσιοποίηση, όταν ζητάει κανείς ε, δημοσιοποίηση, ουσιαστικά πρέπει να έχει διεφαρμόσει το ποσοστό της μόχλευσης, την, αλλογία της μόχλευσης. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ε, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω, γιατί όταν εφαρμόζουμε ένα σύστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και το θέτουμε σε νομοθεσία, δεν φοβάμαι τόσο πολύ αυτούς τους ε, μάνατζερ που μετακινούνται από τις ΗΠΑ, της Σιγκαπούρη και παραπέρα. Όταν ε, δεν μπορούν ε, να πάρουν κάτι παραπάνω από τις αμοιβέ. Μια παραπάνω αμοιβή, δηλαδή ένα σταθερό ποσό μεταβλητής. Ε, εντάξει, αν δεν παίρνουν την αμοιβή αυτή, για μένα μπορούν να φύγουν από την Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει και με το ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη. Εγώ είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής Αναρμόνησης, αλλά θα πρέπει να το καθορίσουμε αυτό και με σαφήνεια για μια πρόσθετη αμοιβή που θα ποικίλει, μεταβλητή αμοιβή. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε και το πώς ε, θα σέβονται αυτή η νομοθεσία την ΕΜΗΡ έτσι λοιπόν, ε, έχω βάλει μια τροπολογία σε σχέση με, τα παράγω, με τις παράγωγες συμβάσεις. Εκεί δεν θα πρέπει να πάμε πέρα από την ΕΜΗΡ, ε, δεν, θα πρέπει και να αποδυναμώνουμε τα όσα έχουμε πετύχει εκεί. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ε, συνέπεια με την εφαρμογή σε τρίτες χώρες. Εγώ συμφωνώ με τις ανησυχίες άλλων συναδέλφων και πρέπει να το διαρευνήσουμε και αυτό αλλά ε, δεν θα πρέπει ε, να αποδυναμώσουμε το κείμενο σε σχέση με την ταχύτητα. Ευχαριστώ κύριο Ζήμπον για τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης που μίλησαν και πολλοί συνάδελφοι θα περιοριστώ σε τρία σημαντικά ζητήματα. Συμφωνώ με τον εισηγητή και πολλούς συναδέλφους πως ε, η πίστοση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ε, καθώς αυτές έχουν μεγάλη σημασία για την ε, οικονομία μας, δεν θα πρέπει να γίνει δυσκολότερη μέσω των υψηλότερων κεφαλαίων απαιτήσεων κατόπιν. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση σε δύο στάδια στην συζήτηση θα μπορούσαν παραδείγματο χάρη να δούμε τι πιστώσει σε φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι το τωρινό πλαφόν του ενός εκατομμυρίου να τις αξιολογήσουμε με το 50% και μέχρι το ύψος των 5 ε, εκατομμυρίων να μειωθεί από 100% σε 75% η στάθμιση του κινδύνου και έτσι θα μειωθεί νομίζω ο κίνδυνος ε, χρεοκοπίας και θα έχουμε υψηλότερο αριθμό δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό είναι η στάθμιση κινδύνου για τα ακίνητα, τις κατοικίες και τα εμπορικά ακίνητα, γιατί η Κομισιόν ζητάει μια αύξηση από 35% σε 50% για τα δάνεια αυτά, κάτι το οποίο σημαίνει πως λόγω της διαφορετικής ανάπτυξης των αγορών ακινήτων σε κράτη-μέλη μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη αυστηροποίηση. Επίσης, ε, στις ε, τωρινές προτάσεις δεν προέπεται μείωση της ε, στάθμισης του κινδύνου για τις ανεπτυγμένες αγορές ακινήτων. Θεωρώ πως η ευελιξία αυτή που υπάρχει για τα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί στο σημείο αυτό. Τέλος, να αναφερθώ στο ποσοστό ε, χρεών. Αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να μελετάμε τις ε, επιπτώσεις ειδικά όταν μιλάμε για μικρομεσαίες τράπεζες που δεν έχουν αναλάβει μεγάλους κινδύνους θα μπορούσε αυτό να έχει μοιραίες συνέπειες για τον ε, όγκο των συναλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν να το ερευνήσουμε. Ένα ενιαίο ποσοστό δικαιολογείται για όλες τις τράπεζες ή θα πρέπει να διαφέρει ανάμεσα με το μέγεθος, ανάλογα με το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο της, ε, κάθε, ε, της κάθε τράπεζας. ανάλογα επίσης και με τις δομές χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης κάθε τράπεζας. Τι αποτέλεσμα είχε επίσης στον ισολογισμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικά αν σκεφτούμε τη χρηματοδότηση δήμων και άλλες επενδύσεις χαμηλού ρίσκου. Και επίσης, και εδώ πέρα θα κλείσω, θα πρέπει να υπάρξει μια δημοσίευση αυτού του λόγου μετά από την απαραίτητη στάθμευση και όχι στη φάση της παρατήρησης γιατί ακριβώς τότε η συγκρισιμότητα θα προκύψει στο τέλος. Κύριε Κάρας, θέλω να σας συγχαρώ για τη δουλειά που έχετε κάνει και εύχομαι καλή δύναμη για αυτά που σας περιμένουν. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στους φιλελευθέρους τώρα. Σίλβια, σε συντονίστρια, μήπως θες να πάρεις πρώτα το λόγο. Thank you, Sharon. No, merci bien. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Οτμάρ. Ε, πολλά υπόθηκαν. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω, σε δύο-τρία σημεία. Καταρχήν, υπάρχει μια παγίδα σε όλα αυτά τα τεράστια πακέτα νομοθεσία που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, χανόμαστε τόσο στι τεχνικέ λεπτομέρειε και ξεχνάμε ποιε είναι οι πολιτικέ επιλογέ. Εμπιστεύομαι τον Οτμαρ για να βρει την ισορροπία αλλά από την πλευρά των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων υπήρχε έγκριση των συμφωνιών της Βασίλειας, αλλά η... στις δημοκρατίες η νομοθεσία γίνεται στα κοινοβούλια. Ε, και παραδείγματος χάρη για το θέμα του ορθού μέτρου μεταξύ της ενίσχυσης της ε, ασφάλειας ε, και του ότι δεν θα επιδεινώσουμε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση νομίζω ότι εξελίχθηκαν τα πράγματα και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Γι' αυτό το λόγο εγώ δεν είμαι υπέρ στο να προτρέχουμε στον τομέα των ΣΥΦΙΣ για το τι πρέπει να γίνει συστημικά ιδρύματα αλλά πολλές φορές βλέπουμε να προτρέχουν οι αλλά και ο ίδιο ο κλάδο, και εγώ δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλό ο αυτό. αυτός. Δεύτερο στοιχείο, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία για μένα και το επενθύμησε και η Κορίν, εμείς ε, ψηφίσαμε ένα πακέτο εποπτείας, δημιουργήθηκαν ευρωπαϊκές οντότητες ε, και εδώ και χρόνια ε, βλέπουμε ότι υπήρχε μία απουσία εποπτείας ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πληρώσαμε το τίμημα. Δεχτήκαμε την αρχή του Single Rule Book, των εγχειριδίου κανόνων και θέλαμε να έχουμε ευρωπαϊκή επιπτωτική ποία για να επιτρέψουμε μια ακόμη φορά για να να επιτρέψουμε στις οικονομικές υπηρεσίες ε, να επωφεληθούν από την η αγορά. Νομίζω ότι κάθε προσπάθεια ε, κράτους να ε, διατηρήσει μικρές εθνικές εξουσίες πρέπει να βρει αντίσταση από εμά και αυτό πρέπει να αποσαφινιστεί από το Κοινοβούλιο μετά την υιοθέτηση της νομοθεσίας για την εποπτεία και φυσικά και στο εσωτερικό των ενχειριδιού κανόνων αλλά και στο επίπεδο 2 μπορούμε να φανταστούμε ε, κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, περιορισμένες ε, αλλά όχι παρεκκλήσεις που θα γίνονται στις εθνικές εποπτικές αρχές αλευκή επιταγή. Νομίζω ότι εδώ ε, διακυβεύεται η εσωτερική αγορά και πραγματικά Βίκη όταν είπες markets ε, στον πληθυντικό εξεπλάγει να έχουμε δικαίωμα στις αγορές, ε, στις δικαιοδοσίες, στον πληθυντικό. Εγώ είχα μάθει ότι μιλήσαμε γεννή αγορά, στον ενικό. Και κάτι τελευταίο επί το οποίο έκανα κάποιες τροπολογίες. Ναι, θα δούμε μια μέρα ε, ε υπερασπίζονται καλύτερα οι Γάλλοι από τους Βρετανούς στην ίδια αγορά, θα γελάσουμε. Να δούμε τώρα τι θα κάνουμε αν δεν υπάρχει εφαρμογή. Ε, δεν θέλω να υποψιαστώ τους Αμερικανούς ή τους Κινέζους ότι δεν θα εφαρμόσουν την νομοθεσία, αλλά βγαίνουμε από μια κρίση και για 10 χρόνια στην Ευρωζώνη ε, Πιστεύαμε ότι αρκούσε να έχουμε κανόνε για να γίνονται σεβαστοί. Ήταν πραγματικό ανέκδοτο αυτό. Και τώρα δεν ξέρω αν έχω τη λύση, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι από κοινού στο τι θα κάνουμε αν δεν εφαρμοστούν οι κανόνε. Τώρα εδώ βρισκόμαστε στην αυτορύθμιση των κρατών. Θα πιστέψουμε εντελώ εννοείται ότι όλοι θα σεβαστούν του κανόνε επειδή κάποια στιγμή υιοθετήθηκαν. Αυτό είναι εντελώ ε, αγαθό, ανόητο. Έτσι λοιπόν, όταν σε ένα μηχανισμό διασφάλιση, ε, κάποια στιγμή ε, μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Ε, αλλά όπως και να έχει ιδέα ότι δεν υπάρχει enforcement, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να επαληθεύσουμε τι οι άλλοι έχουν θέσει σε εφαρμογή ε, και εμείς αμοιβαία αν οι άλλοι έχουν κάποιες εμφιβολίες ε, να τις διασκεδάσουμε. Νομίζω ότι αυτό, το ότι δεν το προβλέπουμε, αφήνει μια τεράστια τρύπα στο σύστημα. Πάντως, έχουμε κατά νου τους στρατηγικούς προσανατολισμούς αυτού του κειμένου και αντί να χανόμαστε σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξαναπερνάμε στο ΕΛΚ. έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον συγγητή που έφυγα, αλλά έπρεπε να ψηφίσω στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Και καταλαβαίνετε, πρέπει ε, και σε εκείνη την Επιτροπή να ρυθμιστούν κάποια θέματα για αυτό που ουσίασα. Θα περιοριστώ σε, σε δύο-τρία ουσιαστικά σημεία που αφορούν και τις τροπολογίες μου σε ό,τι αφορά τώρα την ε, βραχυπρόθεσμη ρεστότητα, liquidity coverage ratio, το άρθρο 413.1. Ε, το να περιορίσουμε τις εισρωές στο 75% σε σχέση με τις εκροές. Αυτός ο μηχανισμός υποχρεώνει τις τράπεζες ε, σε κάθε περίπτωση να κρατούν ένα αποθεματικό ε, ρευστών διαθεσίμων της τάξης του 25% των εκροών ρευστότητας. Ένα τέτοιο σύστημα εφαρμόζεται με ομοιόμορφη όμορφο τρόπο σε όλες τις τράπεζες ανεξαρτήτως της κατάστασης ρευστότητάς τους. Ο περιορισμός του 75% υπάρχει στη Συμφωνία Βασιλεία 3 που εμείς μεταφέρουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μέσω αυτού του νομοθετικού πακέτου CRD4 αλλά στο ε, στην Βασιλεία 3 αυτός ο, περιορισμός αφορά μόνο το πάγιο, το πάγιο επίπεδο, δηλαδή ε, μιλάμε για έναν διασυνοριακό τραπεζικό μήλο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο το ότι εμείς εφαρμόζουμε τους κανόνες προληπτικής επίπεδας και ε, σε μονομή επίπεδο και σε ενωπημένο επίπεδο αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται και ε, σε ενοποιημένο επίπεδο αλλά και σε επίπεδο θρικατρικών ενός ομίλου που την χάνουν προληπτικής εποπτείας μεμονωμένης. Έτσι λοιπόν ε, το σύνολο των θηγατρικών ενό ομίλου θα πρέπει να έχει ένα αποθεματικό ρευστό διαθεσίμων και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμπλοκή ενό τμήματο ρευστότητα, μια ομάδα σε επίπεδο ακόμη και αν, ε, έτσι πληρούνται, αν αυτή πληρούν τα κριτήρια του λόγου ρευστότητα. Ε, δεν είναι κατάλληλο κατά γνώμη μου να δημιουργήσουμε τέτοια αποθεματικά ρευστότητα τεχνητά όταν ε, η χρηματοοικονομική κατάσταση ενός ομίλου είναι υγιής και αυτός ο όμιλος σέβεται το σύνολο των προληπτικών κανόνων φερεγγιότητας και ρευστότητας που προβλέπονται από το 44. Γι' αυτό εγώ προτείνω να καταργηθεί ο περιορισμός στο 75%, το αριθμό του 75% μόνο σε μεμονωμένο επίπεδο και να το διατηρήσουμε σε ενοποιημένο επίπεδο. Αυτό αποτελεί ένα συμβιβασμό ελπίζω αποδεκτό για όλους γιατί θα σεβόμασταν την ε, Συμφωνία της Βασιλείας 3 λαμβάνοντας υπόψη και τις ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες που μας οδηγούν στο να εφαρμόσουμε τους προληπτικούς κανόνες σε δύο επίπεδα, και σε μονομένο και σε ενωπημένο επίπεδο. Φοβάμαι από την άλλη ότι, ένα, ότι κάποια σημεία πηγαίνουν ε, πολύ μακριά σε ό,τι αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων δεν συμφωνώ με του όρου του άρθρου 408.3 που προσδίδει στην EBA την εντολή να καταρτήσει για τις 30 Ιουνίου 2014 ένα τεχνικό πρότυπο καθορίζοντας τη μεθοδολογία υπολογισμού των νεκρών ε, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες δυνάμει της σημασίας του θέματος αυτού και των μεγάλων ποσών ε, που διακυβεύονται εδώ. Πιστεύω ότι η συναπόφαση είναι η πιο κατάλληλη νομοθετική οδός. Ε, και στο ίδιο μήκο κύματο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να της ανατεθεί η εξουσία να νομοθετεί με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις άρθρο 444 για τις τελικές διατάξεις της αναλογίας ρευστότητας, του λόγου ρευστότητας βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή για τα οριστικά ποσά εκροών και για τις εισροές σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες παθητικών και ενεργητικών στοιχείων και ο οριστικός κατάλογο και για τον οριστικό κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων που είναι επιλέξιμα για το αποθεματικό των ρευστών διαθεσίμων που θα πρέπει να κατέχει η τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εκροές της, τις καθαρές net outflows δυνάμει του στρατηγικού τους χαρακτήρα, θα πρέπει κατά την άποψή μου και εδώ να έχουμε μία διαδικασία συναπόφασης προκειμένου αναθεώρηση του καθεστώτος ε, ε, ε, του, ε, της μεγάλης έκθεσης θα χρειαστεί πολύ μεγάλη δουλειά από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από την Κομισιόν, από τον τραπεζικό κλάδο, από τις Εποπτικέ αρχές, από την EBA, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, καθώς και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο, αν υποθέσουμε ότι η Κομισιόν ε, αποφασίσει να προτείνει νομοθετικό κείμενο. Επίσης πιστεύω ότι η προθεσμία της 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν είναι ρεαλιστική. Αν δούμε το νομοθετικό και ρυθμιστικό χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται ενώπιόν μας, έτσι λοιπόν προτείνω αναβολή της αναθεώρησης του καθεστώτος ε, του Μεγάλου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 την ημερομηνία στην οποία θα έχουμε θέσει σε εφαρμογή το σύνολο του μηχανισμού Βασιλεία 3 CRD4, κεφαλαϊκές απαιτήσεις 4, βάσει και των ε, μεταβατικών περιόδων που θα έχουν προβλεφθεί στον μηχανισμό. Αυτή είναι η εξήγηση τροπολογιών μου, Πρόεδρε, και ελπίζω ότι ο συγητής μπορεί να τις λάβει υπόψη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια ο Γκούναρ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Ότμα Κάρα για εξαιρετική έκθεση, εισήγηση. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές για το πνεύμα συνεργασίας και για τον διάλογο. Είναι εύκολο να δει κανείς αυτή την έκθεση ως τεχνικής μορφής έκθεση, διότι υπάρχουν τεράστιες τεχνικές λεπτομέρειες, πολλές πάμπολες και βλέποντας όμως τη στόχευση του εισηγητή που είναι πολιτικού χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για την σταθεροποίηση και την ικανότητα να βρούμε τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία σε αυτή την αλληλουχία. Για μένα ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η διασφάλιση ότι θα έχουμε υψηλότατο επίπεδο ευθυνών και λογοδοσία στον τραπεζικό τομέα. Και με το ανώτατο αυτό επίπεδο λογοδοσίας και ευθυνών θα είναι αναγκαίο να είναι εφικτό και λειτουργικό αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό και για το corporate governance, την ε, εταιρική διακυβέρνηση ή διαχείριση πρέπει να μπορέσουμε να καταστήσουμε αυτό το πλαίσιο εφικτό για όσους εμπλέκονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής των ε, εταίρων ε, ώστε να επιτευχθεί αυτό. Δεύτερο για την ευθύνη, η εταιρική ευθύνη είναι ότι έχει τεράστια σημασία να έχουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά που θα είναι ανοιχτή και θα λειτουργεί σωστά. Αυτό δεν αποκλείει όμως για εκείνα τα κράτη-μέλη που έχουν διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο τραπεζικός τομέας τους και έχουν διαφορετικά μερίδια, μερίδα στην οικονομία να μπορούν να αναλαμβάνουν διαφορετικές δράσεις όσον αφορά και το υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης μια και έχουν και μεγαλύτερους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ως έσχατη ανάγκη. Ας πάρουμε ένα ε, έσχατο παράδειγμα στον ε, τομέα της ε, Could be quite appropriate that Iceland... την Ισλανδία με τον τραπεζικό τομέα που ε, θα μπορούσε να ενταχθεί στο ε, μεγαλύτερο πλαίσιο ε, ευθύνων και κάλυψης. Όμως αυτό δεν είναι το θέμα το οποίο συζητούμε ακριβώς σήμερα. Σε σχέση με το σχετικά μεγάλο τμήμα στην οικονομία τραπεζικών οργάνων. Θα πρέπει να μην υπάρχει στρέβλωση, να μην υπάρχει υπονόμευση του ανταγωνισμού με τα μέτρα αυτά και να συνεισφέρουμε στην σταθεροποίηση και σταθερότητα στην απάλληψη ή αναχέτηση συστημικών κινδύνων. Και σοφό θα ήταν και συνετό αν ε, μπορούσαμε να δώσουμε την δυνατότητα σε τέτοιες χώρες με τέτοιο μέγεθος ε, τραπεζικών ε, ιδρυμάτων να αντιμετωπίσουν με το σωστό τρόπο τους συστημικούς κινδύνους. Και δεύτερον, τα κάνουμε λόγο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες για το τραπεζικό σύστημα να παρέχει κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η σωστή ισορροπία και η σωστή στάθμιση κινδύνων. Γιατί αν δούμε όλους τους κινδύνους ε, ισοπεδωτικά ως ε, ίδιους και ίσους, ε, τότε αυτό θα αποβεί εις βάρος των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν όμως διασφαλίσουμε ότι θα καλύπτουν με τη σωστή ανάλυση τους ενδεδειγμένους κινδύνους οι τράπεζες, θα υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα με την δυνατότητα σταθεροποίησης και διασφάλισης των επενδύσεων, των δανείων, των πιστώσεων. Σημαντικά θέματα αυτά στην, Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτές τις επιχειρήσεις. Έτσι με ένα λεπτό 54 δευτερόλεπτα ολοκληρώνω και νομίζω αυτό είναι μοναδική επίδοση και αυτό υπογραμμίζει το μέγεθος ε, του μηνύματος που ήθελα να αποστείλω. Σας ευχαριστούμε. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να αναφέρω ότι εδώ γινόταν και παρέμβαση εξ του συναδέλφου. Πώς είπατε Ακριβώς γνωρίζω πόσο, επί πόσο χρόνο ε, παρεμβαίνουν οι συνάδελφοι. 12 σκιώδεις εισηγητές, 20 άλλοι και άλλοι για 6 λεπτά. Είναι μια τέλος πάντων αναλογία δεδομένη αυτή. Επόμενη παρέμβηση, Άντρε Σβάμπ. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, τροπολογίες ε, που είναι πειρασμός να μακρηγορήσει κανείς. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι δεν επιθυμεί να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για διαφορετικές τράπεζες. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο ως προσέγγιση για όλες τις τράπεζες και γι' αυτό έχει την πλήρη υποστήριξή μου. Παρ' όλα αυτά παρόλες τις τροπολογίες και τις δυσκολίες να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς, θέλω δύο σημεία σύντομα να αναφέρω με δικά μου λόγια που είναι σημαντική υπόθεση για την αναζήτηση συμβιβασμών. Πρώτον, έχουμε κάθε συμφέρον θα έλεγα και το λέω και ως εκπρόσωπος ενός κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως εχόντων των πραγμάτων. Η στάθμιση κινδύνων να τηρηθεί στο σημερινό επίπεδο. Αν θα το κάνουμε όπως προτείνει ο συνάδελφος Σίμων ή όπως προτείνεται από τους Πρασίνους ή ακόμα και με μια καλύτερη πρόταση του συναδέλφου Καράς, το αφήνω ανοιχτό. Όμως ο κίνδυνος ε, έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν ήταν ε, το αίτιο της κρίσης ε, και γι' αυτό έχουμε κάθε συμφέρον να τηρήσουμε τα πράγματα σε αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, για τη συμμετοχή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις. Η αυστηροποίηση για τους ε, λόγους που αναφέρονται είναι κάτι κατανοητό βέβαια, αλλά όμως τους μικρομεσαίους ε, θα τους ε, δυσχεράνει και θα τους επιβαρύνει και αυτό το οποίο ανέφερε τώρα μόλις η Astrid Λούλινγκ. Είναι σωστό να μην έχουμε ε, ξεχωριστή αρμοδιότητα για την ΕΜΠΑ, αλλά να έχουμε ε, μια συντονιστική δράση. Δεν έχει μέχρι σήμερα την οριμότητα το ΕΜΠΑ να δράσει στις αγορές ε, και αυτά τα οποία είδαμε κατά τους προηγούμενους μήνες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ίσως τα καταφέρει καλύτερα στο μέλλον, αλλά είναι πρόημο εκείνη να αποφασίζει αποκλειστικά. Σας ευχαριστώ, Άντρεα και ευχαριστώ που είσαστε σύντομος. Ο Αντολίν Σάντσες Πρεθέντο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα, να, συνεισφέρω. συνεισφέρω. Θα ήθελα να συνεισφέρω σε αυτή τη συζήτηση και εγώ, επεξηγώντα ποιο είναι ο προσανατολισμό των τροπολογιών μου, για να μπορέσει να συλλάβει υπόψη ο εισηγητή και σε σχέση με τι διαπραγματεύσει που θα κάνει. Ο στόχος μου είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των δικών μας επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να γίνει με την ενίσχυση της ίδιας ε, της εταιρικής διακυβέρνησης και με την αποφυγή του να επιβαρυνθούν με ιδιαίτερα υπερβολικά βάρη και άχθη που δεν θα τους δώσει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικές. Για την διαχείριση διακυβέρνηση Πρέπει να αποφύγουμε να είμαστε υπερβολικά επεμβατικοί σε σχέση με τις επιχειρήσεις και τις δομές τους. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να διασφαλίσουμε όμως ότι θα υπάρχουν ε, προδιαγραφές τουλάχιστον συγκρίσιμες ε, ώστε με αυτά τα οποία θα ε, θεσπίζουμε να μην υπερβάλλουμε και στρεβλώνουμε ώστε για την διαχείριση του managing body να υπάρχει ένα ε, σωστό πλαίσιο λειτουργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά και την λειτουργία των προδιαγραφών που θα πρέπει στο, ε, στους κόλπους τους να λειτουργούν δεν ήμουν όσον αφορά αυτό το θέμα ε, καινοτόμο, όμω ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση αστοχεύουν. Δεύτερο, για τι ε, αρχέ εποπτεία. Είμαστε σε μια ενιαία εσωτερική αγορά και πρέπει αυτό να είναι σαφέ για όσου εμπλέκονται. Υπάρχουν διαφορέ σε σχέση με κάποιε αγορέ για τον στεγαστικό τομέα, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δούμε τι διαφορέ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τι προποθέσει Τη της ε, αγοράς. Όταν υπάρχουν λοιπόν διαφορές ε, σε σχέση με την χώρα υποδοχής ε, και την επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ως γατρική σε αυτήν, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τις πτυχές της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Και αυτό να μην γίνεται εις βάρος της ρύθμισης ε, που θα βρίσκεται κάτω από το ε, αναγκαίο επίπεδο. Ως προς αυτό θα πρέπει να είμαστε ε, σαφέστατοι. Επίσης πιστεύω για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγούμενα ότι αν θέλουμε να αυξηθεί η αηφορία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δραστήρια της τα αίτια των κυκλικών, της κυκλικής επανάληψης τέτοιων φαινομένων. Και γι' αυτό θα πρέπει η τελική λύση να ε, στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Για τις ε, επενδύσεις ε, όσον αφορά τις θηγατρικές είναι και αυτή μια σημαντική πτυχή. Πρώτον, για να μην υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τις θηγατρικές, όπως π.χ. τον είπα. και γιατί το software και αυτό συνεπάγεται ένα τομέα αποτελεσματικό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε επαρκώς το κεφάλαιο των θηγατρικών, μπορεί να δώσουμε κίνητρα να υπάρχει μια αποσταθεροποίηση και αυτή δεν είναι η σωστή πορεία. Η σωστή πορεία θα ήταν να προσπαθήσουμε σε ένα επαρκέ πλαίσιο να πρικοδοτήσουμε αυτές ε, τις ανάγκες. Και όσον αφορά και τις απώλειες, στην ενιαία εσωτερική αγορά ένα σημαντικό στοιχείο είναι η συγκρισιμότητα, συγκρισιμότητα στοιχείων θα πρέπει να θεσπίσουμε σαφείς μηχανισμούς ώστε οι απώλειες ε, να μπορούν να είναι συγκρίσιμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί διαφορετικά κάθε ένα από τα πρότυπα θα οδηγούσε σε δυσκολίες ε, στο να υπάρξει ένα κοινό πρότυπο και ένα κοινό συγκρίσιμο πλαίσιο. Σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν από πλευρά του εισηγητή για προβλέψεις όσον αφορά το Financial Stability Board να εισαχθούν κάποια στοιχεία σε σχέση με το θέμα αυτών των δανείων. Και στο θέμα της ρευστότητα τέλος θα ήθελα να καταφέρουμε να λάβουμε υπόψη το θέμα των ομολόγων. Να είμαστε σαφείς αυτό το οποίο ε, θέλουμε να αποφύγουμε είναι η τοξική χρήση τέτοιων ομολόγων. Ε, και ένας καλός μηχανισμός πρέπει να εξευρεθεί ώστε σε μια τέτοια σημαντική στιγμή για την ανάκαμψη, την ε, πρόθεση της οικονομίας μας να μην δημιουργήσουμε υπερβολική επιβάρυνση για τέτοιου είδους διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άγγελσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους ε, σκιώδες εισηγητές για την προσέγγιση τους ε, στην ευελιξία. Γιατί εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω, επειδή είμαι και Δανέζα, νομίζω πως το φαντάζεται ο κύριος Κάρας. Το ε, έχω δει και σε έρκέτε τροπολογίε μαζί με άλλους συναδέλφου για τους κανόνε περί ε, και σχετίζεται με την κατάσταση για τα πιστοτικά ιδρύματα ε, που δίνουν στεγαστικά δάνεια. Δύο τρίτα των δανείων περνάνε από αυτά τα πιστοτικά ιδρύματα. Δεν έχουν καταθέσεις, είναι ένα πολύ σταθερό σύστημα που βασίζεται σε μια ισορροπημένη αρχή με ξεκάθαρο κίνδυνο είναι για τους δανειζόμενους χαμηλό κέρδος για τα ίδια τα πιστοτικά ιδρύματα. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες αυτή η ιδέα είναι γιατί δεν δημιουργεί πλούσιους τραπεζίτες. είχε λειτουργήσει σε πολύ δύσκολους ε, καιρούς μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, οπότε είναι ένα εύρωστο σύστημα. Η πρόταση της ε, Κομισιόν και του κυρίου Κάρας οπωσδήποτε αφαίρεσε κάποια προβλήματα της Επιτροπής της ε, Βασιλείας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητήματα για τη ρευστότητα. Δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες. Απλά να πω πως ε, τα ανέφεραν οι παρόντες. Επίσης ε, κάποιες ε, προτάσεις άλλων συναδέλφων θα δημιουργήσουν νέες δυσκολίες. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για την αξιολόγηση των τροπολογίων. το σταθερό αυτό ποσοστό χρηματοδότηση. έχει συζητηθεί και ο κύριος Κάρας είπε να εξετάσουμε τον τρόπο αξιολόγηση και το πώς θα πάει η αξιολόγηση. Ε, κατά την άποψή μου δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, είναι και ζήτημα εξόχως ε, πολιτικό. Και τέλος θα αναφέρω το ζήτημα της Βασιλείας 1 που ανέφερε η Βίκη Φόρντ όπου έχω μαζί με άλλους υποβάλει μία τροπολογία συμβιβαστική η οποία δεν αφαιρεί βεβαίως τη βάση της ε, Βασιλείας 1 αλλά δίνει στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή κάποιες αρμοδιότητες ε, για να αξιολογήσει πότε μπορεί να ισχύσει και πότε όχι. Είναι περισσότερο συμβαστική τροπολογία. Οπότε μένω τις συζητήσεις και το να βρούμε μια καλή και ευέλικτη λύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παύλο. Ευχαριστώ, Σάρων. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σιγητή για το έργο του και για το έργο που θα πρέπει να υλοποιήσει και στο μέλλον που σίγουρα θα είναι αρκετά βαρύς ότι αφορά το δημόσιο κέρδος. Ζούμε ε, κάποιες ε, έκτακτες περιστάσεις και όλοι αγωνιζόμαστε για να μην επαναληφθούν αυτές οι συνθήκες. Έτσι λοιπόν, ε, γι' αυτό εγώ δεν δέχομαι την πρόταση να αυξηθούν οι κεφαλικές απαιτήσει του δημοσίου χρέους. Το δημόσιο χρέος θα πρέπει να είναι ε, κάποιο ελεύθερο διθέσιμο κινδύνου. Διαφορετικά θα θέταμε σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θα δείχναμε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη και στους εαυτούς μας. Επίσης θα δείχναμε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κάνουμε τα απαραίτητα για να διατηρήσουμε την οικονομία μας σταθερή. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να κινηθούμε πολύ προσεκτικά για να μην στείλουμε ένα λανθασμένο μήνυμα σε σχέση με τους εγώ συμφωνώ τόν πρέπει να έχουμε κατά νου τι έχει παραχθεί από τις τράπεζες ε, γιατί πρόκειται για διαθέσιμα που μπορεί να συνεισφέρουν στην πληρωμή ε, των ε, οφειλών σε πιθανή ρευστοποίηση. Επίσης, κάποιες εθνικές νομοθεσίες όπως των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρεί ότι είναι άειλα ε, στοιχεία του ενεργητικού τώρα. Ε, νομίζω ότι ε, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο το να αναγνωρίσουμε για τον όμιλο τις μέγιστες απαιτήσει που απαιτεί η αρχή σε σχέση με τη θηγατρική. Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, θεωρώ ότι το πρωταρχικό είναι η ασφάλεια δικαίου και ε, σύμφωνα με τη δέσμευση των κεντρικών τραπεζών εκεί πρέπει ε, να δούμε ε, ποιες περικοπές εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά τις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Έχουμε καταθέσει μια τροπολογία με ένα διπλό στόχο ο πρώτος στόχος είναι να πετύχουμε μία αύξηση της χρηματοδότησης ε, των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να αποφύγουμε περιορισμό την πίστοση λόγω ε, τέτοιων εκθέσεων ε, βάζοντας πιο λογικές κεφαλαϊκές απαιτήσεις έτσι ώστε τα ιδρύματα να μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και από την άλλη να αυξήσουμε το όριο της κατηγοριοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να αυξήσουμε μειώνοντας το κίνδυνο ε, από 1 εκατομμύριο ευρώ σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Ευχαριστώ Σάρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο ακόμα μιλητέ έχουμε πριν ξαναπάμε στον εισηγητή Χέρμπερτ ε, Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Όσον αφορά την ειδική μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν ήδη. Θεωρώ πως είναι πολύ εξαιρετικός παράγον. Να αναφερθώ τώρα σε κάτι που δεν αναφέρθηκε, την κατάσταση των μικρών συνεταιριστικών τραπεζών σε κάποια κράτη-μέλη και στο δικό μου και στην Ιταλία. Υπάρχει ένα σύστημα με μικρές συνεταιριστικές τράπεζες ε, που μετά ενώνονται σε μεγαλύτερες ε, ε, κοινοπραξίες οι οποίες αποτελούν ένα συνολικό 10% του τραπεζικού τομέα. Θεωρώ πως η ιδιαίτερη κατάσταση αυτών των τραπεζών πρέπει να ληφθεί υπόψη και έχω κάνει σχετικές τροπολογίες σε δύο σημεία. Έχω την 293 για το σύστημα λειτουργίας ε, των συνεταιριστικών τραπεζών. Θεωρώ πως ε, τέτοιοι όμιλοι θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση με άλλους τραπεζικούς ε, ομίλους, δηλαδή την πολλαπλή διοίκηση και δεύτερο θέμα που αφορά πάλι αυτό το σύστημα είναι τα συστήματα διασφάλισης ακριβώς στα συστήματα αυτά στους ομίλους τραπεζών. Υπάρχει μια σύνδεση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην τροπολογία μου υπαριθμών 1159 ε, έχω κάνει μια σχετική πρόταση για τα υπόλοιπα συμφωνώ με όσα ακούστηκαν ευχαριστώ πάρα πολύ Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή Οτμαρ Κάρας για την εξαιρετική δουλειά που έκανε για το ότι επέστησε την προσοχή μας στα προβλήματα τα οποία και εγώ προσπάθησα να αντιμετωπίσω στις τροπολογίες μου. Έχουν ήδη αποσταλεί ε, και θα ήθελα παρόλα αυτά να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχω αποκομίσει την εντύπωση ότι όταν συζητούμε για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει που είναι τόσο σημαντικό ζήτημα για τις αγορές δεδομένων των κινδύνων των αγορών, πολλές φορές συζητάμε για αυτά και δεν συνειδητοποιούμε πάντα το γεγονός ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε την ενιαία εσωτερική αγορά. Είμαι υπέρ της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και φαίνεται ότι και οι Γάλλοι συνάδελφοι όλο και περισσότερο αισθάνονται ότι πρέπει να υποστηριχθεί αυτή η προσέγγιση, αλλά κάνουμε και λόγο για τις ε, υπηρεσίες για αυτήν. Όμως εδώ δεν θα πρέπει να αποσταθεροποιήσουμε το χρηματοοικονομικό σύστημα και ο λόγος είναι ότι το οικονομικό σύστημα υφίσταται και αν προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε, να αλλάξουμε τα ποσοστά ε, ρευστότητας ε, λαμβάνοντας υπόψη τις εταιρείε για τοπικές αγορές που υφίστανται και λειτουργούν κάποιοι κάνουν λόγο για την ε, ε, κοινή αγορά κάποιοι κάνουν λόγο για ε, μερικούς τομείς αυτής της αγοράς πρέπει να προσέξουμε να μην αποσταθεροποιήσουμε αυτό το σύστημα όπως λειτουργεί σήμερα κατά συζήτηση αυτή θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το οποίο προαναφέρθηκε για τις απαιτήσει ε, ποσοτικής μόχλευσης. Πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι τοπικές ιδιομορφίες ε, και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες τοπικά λειτουργούν ε, οι επιχειρήσεις. Και κάνοντας λόγο για αυτές τις ανάγκες πολλά αναφέρθηκαν ήδη προηγούμενα για αυτό το θέμα όμως θα ήθελα να τονίσω ένα θέμα που μάλλον δεν έχει ε, καλυφθεί. Κάνουμε συχνά λόγο για τη Βασιλεία 3, αλλά η Βασιλεία 3 συνιστά ιδιαίτερη σύνεση όσον αφορά ένα πλαίσιο, ένα αρμονισμένο πλαίσιο σύμφωνα με την Βασιλεία 3 οι τοπικές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, και όσον αφορά και τις κεφαλαιακές απο, ε, απαιτήσει. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα προσεκτικοί και σοβαροί για αυτή την υπόθεση. Να έχουμε την δυνατότητα της λειτουργίας της ενιαίας εσωτερικής αγοράς αλλά να μην υπονομεύουμε τα μέτρα ασφάλειας και τις, ε, τα όσα ισχύουν σήμερα και μας προστατεύουν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μια που υπάρχει χρόνος. Ο εισηγητής είπε πως ε, θα ήθελε να ακούσει και την Κομισιόν που βρίσκεται εδώ. Έχετε λοιπόν τον ε, λόγο. Προφανώς ε, μην επεκταθείτε πολύ. Πείτε μας τα, τα βασικά, όχι κάθε τροπολογία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ πλούσια συζήτηση. Δεν έχουμε τη φιλοδοξία να καλύψουμε τα πάντα. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον συγητή και την ομάδα του για την πολύ καλή δουλειά, για την πρόταση αυτή. Είναι εντυπωσιακή η δουλειά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον ε, δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολλέ τροπολογίε και είναι πολύ πλούσια συζήτηση και έχουμε μακρύ δάμο μπροστά μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Άκουσα πολλούς από εσά να επιβεβαιώνετε πόσο σημαντικό είναι γρήγορα να εξετάσουμε το φάκελο, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε και υψηλό βαθμό ποιότητα, επίπεδο ποιότητα. Καλωσορίζουμε και τι δύο φιλοδοξίε φυσικά. Ο κύριος Λαμπέτ είπε ότι ήθελε να ξεκινήσει ανταγωνισμό με το Συμβούλιο <laughs> για να είναι πρώτος. Καλή τύχη σας εύχομαι, γιατί το Συμβούλιο είναι επίσης φιλόδοξο και θέλει να καταλήξει σε συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Έτσι λοιπόν καλωσορίζουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας και στους δύο θεσμούς, ό,τι αφορά τις μικρές και μισές επιχειρήσεις. Πολλοί, αν όχι όλοι, τονίσατε το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σωστή μεταχείριση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Συμφωνεί και η Κομισιόν Έχουμε ε, εντοπίσει το θέμα αυτό από την αρχή ως ένα από τα κύρια θέματα στο όλο εγχείρημα. Θέσαμε και μία ρήτρη αναθεώρησης στην ε, κατάλληλη χρονική στιγμή και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, να κάνει μια ρητρη αναθεώρηση στην καταλληλη χρονικη στιγμη και αξιολόγηση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012. Έτσι λοιπόν φυσικά και εμεί θέλουμε να έχουμε ορθή μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ταυτόχρονα θέλουμε να σα παροτρύνουμε να είμαστε σόφρονε. Δεν ε, πρέπει να προστρέξουμε προς την κατεύθυνση πιο ευνοϊκής μεταχείρισης χωρίς ε, να εξετάσουμε τα απαραίτητα δεδομένα και φυσικά δεν θα ήμασταν αντίθετοι στο να έχουμε τη ρήτρα μάλλον στο, να βάλουμε λίγο πιο μπροστά αυτή τη ρήτρα αναθεώρησης, αλλά θέλουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία, ήδη από σήμερα για να αλλάξουμε το σύστημα ουσιαστικά. Σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ, αυτό υπόθηκε από αρκετούς από εσά. Πολλοί είπατε ότι μπορεί να θέλουμε να είμαστε πιο αυστηροί στο θέμα της αμοιβή και να βάλουμε μία πιο καθορισμένη σχέση μεταξύ του μεταβλητού τμήματος και του σταθερού τμήματος. Ο κύριος Μπερνιέ είπε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και ότι αν οι διατάξεις που εισαχθούν στην πρόταση σε 3 εφαρμοστούν ε, και εφαρμόζονται ήδη από τώρα δεν ε, θεωρηθούν επαρκείς και δεν εφαρμοστούν στην πραγματικότητα, θα ήταν ανοιχτό ε, να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση του συστήματος. Έτσι λοιπόν είμαστε φυσικά έτοιμοι να εξετάσουμε μαζί σας έναν αριθμό πιθανών βελτιώσεων στις διατάξεις περί αμοιβής. Τώρα για τι Ηνωμένες Πολιτείες ή για του άλλου διεθνούς μα εταίρους, και το αν θα εφαρμόσουν τη Βασιλεία 3. Και πάλι εδώ μια βασική ανησυχία για πολλούς από εσά και φυσικά και για την Κομισιόν ε, είναι αυτή. Αναφέρθηκε το πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθεί η κατάσταση και ε, ζητήθηκαν και πληροφορίες από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Από τον κύριο Καρέσα, όπως είπαμε και στο παρελθόν, ε, είπαμε ότι το παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό και σε κάθε περίσταση και ερχόμαστε και είμαστε σε επαφή και με τις ΗΠΑ αλλά και με άλλες δικαιοδοσίες ε, παγκοσμίως. Οι ΗΠΑ ε, τώρα είναι όλο ένα και πιο κοντά στο να εκπονήσουν ένα σχέδιο κανόνων. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Αν ε, σεβαστούν όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα και αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα είμαστε σε θέση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να αξιολογήσουμε πολύ πιο προσεκτικά τι σκοπεύουν να κάνουν ιδέως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε και εμείς να ξεχάσουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Και κάτι ακόμα γι' αυτό, όπως μπορεί να ξέρετε, υπάρχει μια πλήρης διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής στο επίπεδο Βασιλείας. Αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει ήδη. Η Κομισιόν θα συνεισφέρει πολύ στενά και φυσικά και άλλες δικαιοδοσίες ε, θα πιεστούν ε, για να σεβαστούν τις προθεσμίες και να δώσουν και τις απαραίτητες ε, πληροφορίες στην Επιτροπή της Βασιλείας. Και κάτι τελευταίο, αλλά φυσικά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς ενδιαφέρεστε ε, σε αυτό την αναλογία στο επίπεδο 2 και στο εγχειρίδιο κοινών κανόνων. Ε, πολλοί από εσά εκφράσατε υποστήριξη για το εγχειρίδιο κοινών κανόνων και για τη μέγιστη εναρμόνιση, αλλά ταυτόχρονα ζητήσατε και κάποια ευελιξία. Όπως ξέρετε, η Κομισιόν στην πρόταση είχε εισαγάγει μία σειρά εργαλείων ευελιξίας Θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν σωστό και ότι είχε εξευρεθεί κατάλληλη ισορροπία από τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Κατανοούμε ότι το σύστημα μπορεί να χρήζει βελτιώσεων. Σίγουρα θα είμαστε ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο. Όπως και πολλοί από σας είπατε και πάλι σήμερα, πιστεύουμε σε μεγάλο βαθμό στην Κομισιόν ότι αυτό πρέπει να γίνει με ένα πολύ προσεκτικό και ισορροπημένο τρόπο. Έτσι λοιπόν, περαιτέρω ευελιξία για καθορισμένα θέματα ναι, αλλά όχι ει βάρο τη ενιαία αγοράς. Και φυσικά, προς αυτή την κατεύθυνση θα υποστηρίζαμε περαιτέρω συμμετοχή των ευρωπαϊκών φορέων, όπως το ESRB και το MBA, e όπως πολύ προτείνατε. Παρ' όλα αυτά, θα, στο, θα επιμένουμε στο να έχουμε ένα σημαντικό ρόλο παρέμβασης ε, από την πλευρά της Κομισιόν. Έτσι όπως ε, αναφέρθηκε από κάποιους ε, από εσά. Γιατί η Κομισιόν έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ορθής ισορροπίας. Και εδώ θα κλείσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τέλος, για να ολοκληρώσουμε ξανά ο εισηγητής Ότμαρ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, έντονη αυτή και βάθος συζήτηση. Θεωρώ πως μπορώ να πω πως κάποιες παρεμβάσεις επανέλαβαν αυτά τα οποία κατατέθηκαν και συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά και σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη το ότι έχει αλλάξει αυτά, πολλά από αυτά τα οποία α, υπόθηκαν τα αντιλαμβάνουμε ως κάποια έμφαση που θέλατε να δώσετε γιατί πολλά πράγματα που υπάρχουν στην έκθεση αυτή ανταποκρίνονται σε αυτές τις επιθυμίες. Ο κύριος Σβάμπ έχει φύγει αλλά παραδείγματος χάρη για την μείωση της στάθμισης του κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει πρόταση για να μειωθεί κατά 30%. Νομίζω πως είναι ένα θαραλέο βήμα. Δεν ανάγκη να λέμε πως όλα είναι πολύ λίγα και δεν μας ε, φτάνουν. Εάν περάσουμε το 30% νομίζω πως έχουμε κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την ελάφρυνση, την διευκόλυνση των πιστώσεων στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δε αύξηση άλλων ορίων είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εξετάζεται. Και νομίζω πως επιτυχάνουμε περισσότερα με τη μείωση της ε, στάθμισης. Και και μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν ως συμπλήρωμα. Να πω επίσης πως ε, στην Κομισιόν θέλουμε να έχουμε την έκθεση εντός της νομοθετικής διαδικασίας ο Δεκέμβριος 2012 είναι μετά τη λήξη της νομοθετικής διαδικασίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα εντός της νομοθετικής διαδικασίας. Αλλιώς θα το διαπιστώσουμε. Και υπάρχει χρόνος επαρκής κατόπιν για την Κομισιόν ζητώ να ξεκαθαρίσετε πως το Κοινοβούλιο ε, θεωρώ πως εργάζεται εδώ πέρα με περισσότερο θάρρος ε, από ότι το Συμβούλιο και δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την ουδετερότητα στις ε, διαπραγματεύσεις. Θεωρώ πως κάνουμε μια σωστή και καλή πρόταση και δεν νομίζω να αντίθεσε κινδυνός η εφαρμογή. Για το θέμα των ε, συνεταιριστικών τραπεζών ε, και της σχετικής ευθύνης, όλα αυτά υπάρχουν στην έκθεση. Και τον αποκεντρωμένο τομέα και την κοινή ευθύνη και τις συνεταιριστικές τράπεζες και τα ταμιευτήρια όλα αυτά έχουν αναγνωριστεί πλήρως. Είναι ένα μεγάλο βήμα από τη Βασιλεία στην πρόταση της Κομισιόν και στην ε, πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου πως δεν κάνουμε τα πάντα ίδια αλλά λαμβάνουμε υπόψη τις ε, διαφορές αλλά και την ιδιαιτερότητα μεγάλων και μικρών για το ζήτημα του αποκεντρωμένου τομέα των ενώσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το θέμα της κοινή ευθύνη. Όλα αυτά υπάρχουν στις προτάσεις μας και το ότι μιλάμε για την ε, εταιρική δίκηση και εκεί πέρα εξακολουθεί να υπάρχει ο διαχωρισμός με την ε, καθημερινή διοίκηση. Είναι ζήτημα διαφάνειας και διάκρισης των εξουσιών, το λέμε και στην έκθεση Φερέιρα. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει αλλού. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από βάθος καρδίας. Νομίζω πως προχωρήσαμε αρκετά και οπωσδήποτε όταν μπούμε και στις ε, λεπτομέρειες ε, με βάση τις ε, τροπολογίες και τις συμβαστικές προτάσεις σας παρακαλώ να επιδείξουμε ένα πνεύμα συνεργασίας για να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και εμείς δεν θεωρούμε πως υπάρχει εδώ πέρα επίσης κάποια αντίφαση. Το ένα νομίζω θα φέρει το άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να αγνοηθεί ή να θα αγνοείται η Επιτροπή μας από το Συμβούλιο Φεξής. Εντάξει, έχουμε μια άλλη ανταλλαγή απόψε στις 12 Απριλίου, όπου θα έχουμε και άλλες συμβαστικές τροπολογίες που θα πρέπει να καλυφθούν και στοχεύουμε στις 25-26 Απριλίου από πλευράς ε, Επιτροπής μας να τα καλύψουμε. Καταφέραμε να τελειώσουμε τις εργασίες μας νωρίτερα. Κάποιοι θα πάνε για κάποιο καφέ τώρα στο διάλειμμα αυτό. Προειδοποιώ τα μέλη για το απόγευμα όταν θα ακολουθήσει η συνάντηση με την Τρόικα και θα έχουμε και την Επιτροπή Απασχόλησης που θα προσέλθει κατά τη διάρκεια του μεσημερινού διαλύματος θα αλλάξουν οι θέσεις σας. Αν θέλετε να πάρετε τα χαρτιά σας ή τα έγγραφά σας και τα προσωπικά σας αντικείμενα, μην τα αφήσετε εκεί που βρίσκονται, γιατί μπορεί να μετακινηθούν και θα δημιουργηθεί σύγχυση. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Το απόγευμα θα έχουμε συνάντηση συντονιστών στις 3. Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα ξεκινήσουν στις 4. Ευχαριστώ. Γεια.